So, Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με χαρά σας καλωσορίζω στην απογευματινή συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω το τι έγινε με τους συντονιστές Οι συντονιστές ε, σημείωσαν την καινούργια για διάταξη για τη συνεδρίαση 10 και 11 Ιουλίου και συμφώνησαν να εφαρμόσουν την διαδικασία του κατεπήγοντος στην αναφορά 578 του 17 κατόπιν για τις εκθέσεις και τις χρηματοδοτήσεις. Οι σοσιαλδημοκράτες ε, τελικά δεν θέλουν την ε, έκθεση για την στρατηγική για την αναπηρία και, θα το... και το e θα συντάξει την ετήσια έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για τις συστάσεις εγκρίθηκαν ε, και τα τρία αιτήματα για τα σημεία Β τα οποία θα περιληφθούν ε, στα γραπτά πρακτικά. Επίσης ε, συζητήθηκε το θέμα των ε, επισκέψεων των διερευνητικών, η επίσκεψη των Τάραντα. Συμφωνήσαμε για το πρόγραμμα, κατόπιν έχουμε την επίσκεψη στη Λάρνακα το Σεπτέμβριο. Και μετά συζητήσαμε την επίσκεψη στην Ισπανία είχα μια πρώτη ενδιαφέρουσα συζήτηση αλλά τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα και υπάρχει επίσης μια ξεκάθαρη απόφαση για τις ακροάσεις για τους απάτριδες πότε είναι 29 Ιουνίου μάλιστα Επίσης οι συντονιστές ε, συμφώνησαν για το τι θα γίνει με την αναφορά 747 του 2016 όπως επίσης ε, και το σχέδιο ενσωμάτωσης της πολιτικής ε, του φίλου αλλά και το αίτημα του ΙΕΝΕΦ για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, προσωρινών εργαζομένων. Και βέβαια ενημερώσαμε και για το τι έγινε στην διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών στις 7 και 13 Ιουνίου. Αυτά λοιπόν και τώρα θα δώσω τον λόγο για την συζήτησή μας για τις νέες αναφορές. Έχουμε την αναφορά 164 του 2017. Συντάκτης είναι κ. Σλόιντ από τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον αναφέροντα. Καλώς ήρθατε, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και για την πρόσκληση. Αν μου επιτρέπετε να σας δώσω κάποιες ε, λεπτομέρειες ε, για μένα. Ε, Πρώτη μου αναφορά Ήμουν η πρώτη που κατέθεσα αναφορά το 1977 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μία ομάδα γυναικών από το Κάρντιφ ε, στην Ουαλία ήταν με ένα μίνιμπας με μία αναφορά και ζητούσαμε ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και μας χαιρέτησαν με μεγάλο ενθουσιασμό γιατί ήμασταν οι πρώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και πολλές ε, φίλες μου ήξεραν ότι ε, τους αναφέρτες. Και όταν έγινα ευρωβουλευτής το 1979 ήμουν πρώτα μέλος της Επιτροπής ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και κάποια τα νομοθετήματα που ζητούσαμε το 1975 εγκρίθηκαν κατόπιν ως ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχω κάποιο ιστορικό θα έλεγα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ε, πετύχαμε κάποια πράγματα από αυτά τα οποία θέλαμε. Πέρασα πέντε χρόνια εδώ ναι, εξελέγει με πρόγραμμα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί το καιρό εκείνο το κόμμα μου ήταν διχασμένο, η μισοί στήριζαν την Ένωση, οι άλλοι μισοί ήταν εναντίον. Εγώ κατεβήκα με πρόγραμμα ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μετά από δύο χρόνια άλλαξα άποψη και θα ήθελα να τονίσω πως ε, είναι καλό να αλλάζει κανείς γνώμη αν ε, δει κάτι που τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Αυτό ισχύει γενικώ. Και έμπλεξα βεβαίως γιατί το ότι η Αγατική ήταν διχασμένη η μισή ήταν υπέρ, η άλλη μισή ήταν κατά οπότε θυμάμαι ότι είχα γράψει ένα άρθρο στο New Statesman και εξηγούσα γιατί άλλαξα άποψη και ένας συνάδελφό μου ήρθε στο διάδρομο και με έδειχνε και έλεγε «Εσύ, εσύ έχασες, εσύ μας έχασες την έδρα του Hillhead» ε, λόγω του άρθρου αυτού και γέλασα εγώ και είπα «Πόσοι διαβάζουν στη Γλασκόβη, στο Hillhead, το New Statesman» δεν είπε τίποτα και μου κόψε την καλημέρα για δύο χρόνια. Ήταν λοιπόν τεταμένη η κατάσταση, πολλωμένη θα έλεγα. Όταν τότε ήμασταν λοιπόν κατά της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ε, τότε βεβαίως μιλούσαμε για βουνά από βούτυρο και λίμνες από κρασί και όλα αυτά τα οποία χρηματοδοτούσε η κοινή γεωργική πολιτική χρόνια πριν από την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου που περιέλαβε νομοθεσία για την ισότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν υπήρχε πολιτική για το περιβάλλον, αλλά μετά από πολλά χρόνια συνεργασίες με συναδέλφους από όλες τις χώρες ειδικά στην σοσιαλιστική ομάδα εργαστήκαμε για τις πολιτικές που όλοι θέλαμε να περάσουμε. Θεωρώ λοιπόν πως υπάρχει όφελος στην συνεργασία με ανθρώπους από άλλες χώρες για ένα καλύτερο μέλλον, για τις δουλειές, για την ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, από το 79 μέχρι το 84 ήμουν ευρωβουλευτής ε, και είδα πως ε, απέκτησε περισσότερες αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο όπως και έπρεπε και προς δυσφορία των Εθνικών Κοινοβουλίων και τώρα έχει τρομερές εξουσίες και αρμοδιότητες και ε, το υπενθύμησα και στην Πρωθυπουργό μας ε, προσφάτως, στην Τερέζα Μέη, στην Βουλή των Κοινοτήτων, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το πάρει πολύ στα σοβαρά στις διαπραγματεύσεις. Και ειδικά βεβαίως έχει στο τέλος ε, την δυνατότητα να προβάλλει βέτο. Και όλοι ξέρουμε από τον ΟΗΕ πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και βεβαίως δεν λέω ότι θα φτάσουμε ως εκεί. Αλλά είναι μια εξουσία την οποία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε. Υπενθύμησα. Το υπενθύμησα λοιπόν στην Τερέζα Μέη. Είπα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό και θα κρίνει την τελική συμφωνία απόσυρσης ε, παρά το ότι δεν έχει επίσημο ρόλο στην διαδικασία του Brexit εκτός από το δικαίωμα να ενημερώνεται. Αλλά θα πρέπει να δώσει την σύμφωνη γνώμη του με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων ε, μελών πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία απόσυρσης. Οπότε το δικαίωμα του Ηνωμένου Βασιλείου να μην κυρώσει την τελική συμφωνία του δίνει ε, σημαντική αρμοδιότητα, ουσιαστικά βέτο. Η αναφορά μου δεν ξέρω, φαντάζομαι την έχετε διαβάσει όλοι. Ναι, ασχολείται με τρεις συγκεκριμένες ανησυχίες από τη συνθήκη της Λισαβόνας, άρθρο 10, παράγραφη 1 και 3, που λέει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Εγώ λοιπόν λέω ότι βεβαίως ε, θα προστατεύσετε τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που εργάζονται στον Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως. Θα σκεφτείτε το πώς θα, επιστρε... επιτρέψετε στους Βρετανούς πολίτες να εργαστούν όταν ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις και βεβαίως ε, θα συζητήσετε κάποια από αυτά τα ζητήματα για να επηρεάσετε το Συμβούλιο και την Κομισιόν έτσι ώστε να έχουν αυτά τα ζητήματα σε υψηλή προτεραιότητα στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Και επίσης προτείνω στην αναφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσκαλέσει την Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα και να απαντήσει ερωτήσεις για ε, ε, τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία. Τα έχω πει αυτά ήδη και στην ε, Τερέζα Μεή, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και την ρώτησα εάν θα εμφανιζόταν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να απαντήσει ερωτήσεις και η απάντησή της ήταν ότι δεν είχε λάβει κάποια πρόσκληση αλλά αν ελάμβανε θα το σκεφτόταν πολύ προσεκτικά. Είδω λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί κάποια συνέχεια. Γιατί έχω παρακολουθήσει κάποιες από τις συζητήσεις σας και νομίζω ότι φύγεται κάποια σημεία που ανησυχούν και εμάς που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπωσδήποτε οι ψηφοφόροι μας και μόλις είχαμε εκλογές ε, παρά το ότι περισσότεροι στην εκλογική μου περιφέρεια στην Νότια Ουαλία ψήφισαν να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επηρέασε αυτό τα δικά μου εκλογικά αποτελέσματα. Εγώ προφανώ είμαι υπέρ του να μείνουμε στην Ένωση. Δεν με επηρέασε λοιπόν καθόλου. Αντιθέτω. Ανέβηκε η πλειοψηφία μου, πήρα 61% των ψήφων. Δεν είχα λοιπόν κάποιο ένα πρόβλημα. με ψηφοφόρου τα δύο τρίτα των οποίων ε, είχαν ψηφίσει διαφορετικά. Λοιπόν, στις εκλογές ε, πήγαινα χτυπούσα πόρτες, μιλούσα με τον κόσμο και τους ανησυχούσε η βιομηχανία την ε, Ford που είναι μεγάλος εργοδότης εκεί είπαν ότι ανησυχούν πολύ για το μέλλον της βιομηχανίας εάν βγούμε από την Ένωση και κάποιος ο οποίος δουλεύει στην Panasonic που και πάλι είναι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία είπε ότι και αυτός ανησυχούσε πολύ. Λοιπόν, είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που είχα ακούσει. Είχα αγοράσει κάτι ηλιοτρόπια από ένα πλανόδιο σε μια λαϊκή αγορά και του μιλούσα δεν τον είχα ξαναδεί και ήταν ένας Ιταλός που έχει ζήσει 15 χρόνια στην Ουαλία και είπε πραγματικά έχω συγχυστεί και του λέω γιατί γιατί μου λένε όλοι τώρα θα, θα φεύγεις σιγά σιγά ε? δεν είναι ώρα να φεύγεις να πηγαίνεις στη χώρα σου και τους λέω μα έχω ζήσει 15 χρόνια εδώ εδώ είναι η χώρα μου και περιμένουν ένας πολίτης της Ένωσης επειδή δεν είναι Βρετανός, να αρχίσει να φεύγει σιγά σιγά. Λοιπόν, ανησυχούν ε, πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που έχουν πολλούς δεσμούς. Ε, άνθρωποι, ε, νοσηλευτές. Βλέπουμε ότι δεν προσλαμβάνουμε σε νοσοκόμες όσο το παρελθόν από το εξωτερικό, γιατί ο κόσμος φοβάται ότι θα τους στείλουν πίσω. Μπορούσα να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά ο πρόεδρος μου κάνει νόημα. By Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι το 2017 ότι είμαστε καλύτερα ενωμένοι. Αυτοί οι οποίοι ε, θα πανηγύριζανε αν φεύγαμε από την Ένωση και μερικοί πολύ αντιπαθητικοί άνθρωποι που τους ξέρετε πολύ καλά εδώ μέσα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται την κλιματική αλλαγή που δεν θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τους πιο ευπαθείς της κοινωνίας μας. Λοιπόν, για την ευμερία, για τη συλλογική ασφάλεια, αν θέλουμε μια οικονομία και μια κοινωνία που θα λειτουργεί για όλους. Ε, εξακολουθώ να θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα εντός της Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. If you allow me, I would like to continue in... Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσω ουγγρικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της αναφοράς, για τα λόγια σας. Ως πρόεδρος της Επιτροπής δεν ε, μπορώ να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, αλλά για μισό λεπτό θα ήθελα εδώ να κάνω μία εξαίρεση. Και να πω ότι υπάρχει ένας μόνο που μπορεί να αλλάξει την ε, απόφαση για τον Brexit και αυτός ο ένας είναι ο Βρετανικός λαός. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν μόνο μπορεί να αντιστρέψει την απόφαση και να αλλάξουν τα ποσοστά του ναι και του όχι. Εσείς μας είπατε πως αλλάξατε άποψη και ίσως ε, αλλάξει και η άποψη των ψηφοφόρων σας και αυτό θα ήταν πολύ ευχάριστο, θα το χαιρέτιζα εάν ξαναγύριζαν κοντά μας οι Βρετανοί. Ανάλαζαν γνώμη το 2018-2019. Αν μπορείτε να αλλάξετε το κλίμα, τότε εμεί θα σας στηρίξουμε. Όμως αυτή είναι μια απόφαση που μπορούν να λάβουν μόνο οι Βρετανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναφορά, θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους και θα πω ότι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως ε, καθήκον να ακούει τους πολίτες, να τους δίνει ένα βήμα, να μιλήσουν, να πούν τη γνώμη τους. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Ακούμε πολλές σκέψεις, πολλούς φόβους, ακριβώς εξαιτία αυτής της απόφασης της Μεγάλης Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι σήμερα δεν μπορούμε να πάρουμε καμία ευχάριστη απόφαση για καμία αναφορά που έχουμε στην μερισία διάταξη ε, λόγω του περιεχομένου της. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή, να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις ανησυχίες του Βρετανικού λαού και να συνοδεύσουμε ε, τους Βρετανούς στη διαδικασία αυτή σε όλη τη διάρκεια. Μέχρι το 2019, αλλά και μετά είμαστε εδώ. Και η πρόσκληση που αναφέρατε προς την Τερέζα Μέη είναι κάτι που σημειώσαμε και θα το μεταφέρουμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Άννη και τα υπόλοιπα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων που στήριξαν αυτή την αναφορά και τα μέλη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι νομίζω ένα σημάδι, ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί πως η Επιτροπή Αναφορών, ε, οι βουλευτές μάλλον, θεωρεί πως η Επιτροπή Αναφορών εδώ είναι ένα βήμα για να ακουστούν, για να ακουστεί η φωνή τους στα θεσμικά όργανα. Και το συγκεκριμένο θέμα που αφορά το διάλογο ανάμεσα στην, ε, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και στους Ευρωβουλευτές είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως ε, πολύ καλώς έγινε παραδεκτή αναφορά και τη συζητάμε εδώ. Είναι πιστεύω κομμάτι της κληρονομιάς που θα αφήσουμε να φέρουμε αυτή την αναφορά από το Ηνωμένο Βασίλειο, να συζητήσουμε και άλλες αναφορές, ε, διότι οι Βρετανοί αυτή τη στιγμή ανησυχούν ε, για το βασικό δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης. Είναι, πιστεύω, σημαντική κληρονομιά για το μέλλον. Με θλίβει βέβαια αυτό και λυπάμαι για αυτό ίσως δεν γνωρίζετε όλοι ε, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ορισμένα μέλη των συντηρητικών που ίσως ε, γνωρίζουν, αλλά σήμερα στο Κοινοβούλιο η Βασίλισσα έκανε μια ομιλία για την ημερήσια θέταξη της μειονοτικής ε, κυβέρνησης. Δεν είπε ούτε μία λέξη για τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτή θα ήταν μια ευκαιρία να συζητηθεί ε, αυτό το θέμα, τα δικαιώματα των πολιτών, να ανοίξει ένα τεράστιο ε, διάλογος, όχι μόνο στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά και στην Βουλή των Λόρδων, να καθυστερήσει η διαδικασία. Διότι υπήρξε πολύ μεγάλη αντίσταση, υπήρξε ε, αντιπολίτευση και από τους εργατικούς και από άλλα κόμματα που προσπαθούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τίποτα όμως δεν συζητήθηκε, τίποτα δεν έχει δρομολογηθεί, δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόταση για το επόμενο έτος και αυτό είναι λυπηρό. Στέλνει ένα πολύ δυσάρεστο μήνυμα για όσους έχουν μείνει μετέωροι τον τελευταίο χρόνο, όσους έχει αφήσει η κυβέρνηση στους. Αυτό είναι κάτι που ε, θα έπρεπε να είχε κάνει η κυβέρνηση μου. Να δώσει δηλαδή κάποιες ε, εγγυήσεις, να καθησυχάσει τους πολίτες. Η αναφορά αυτή έχει τύχει τη στήριξη άλλων ε, μελών, άλλων μελών του Κοινοβουλίου, άλλων βουλευτών, όμω η στάση της ε, κυβέρνηση μου είναι τελείως αντίθετη. Έχασαν, πιστεύω, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τοποθετηθούν, να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών και να δείξουν προοδευτική στάση η ατζέντα του Citizens First στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που τραβά τη, συζήτηση προς τα εκεί, που ζητά να υπάρχει κάποια κοινωνική ασφάλιση για τους πολίτες. Εμείς έχουμε, να σας πω και εδώ στην αίθουσα, έναν εκπρόσωπο της ε, Βουλής των Κοινοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά την αναφέρουσα που μας παρουσίασε την αναφορά της, υποβάλλοντας και κάποιες σκέψεις σχετικά με την απόφαση αυτή μετά το δημοψήφισμα. Μας μίλησε και για κάποιες ιδέες, τέλο πάντων, σχετικά με ανταλλαγές, με και όπως είπατε και εσείς είναι σημαντικό να ακούμε τους αναφέροντες από τη Βρετανία όπως σήμερα το απόγευμα ή και από τις άλλες χώρες. Σήμερα το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να τηρείται. Αυτή είναι η μόνη βεβαιότητα. Κατά τα άλλα, καταλαβαίνω το συνέστημα που προβάλλουν οι Βρετανοί συνάδελφοι στη συζήτηση αυτή και η πλειοψηφία ημών νομίζω ότι είμαστε πολύ στεναχωρημένοι μετά την απόφαση των Βρετανών. Πάντως λυπάμαι που κατά τη διάρκεια για το δημοψήφισμα η φωνή των Ευρωπαίων από τις άλλες χώρες δεν ακούστηκε και πολύ. Θυμάμαι πολύ καλά, ας πούμε, ότι Βρετανοί συνάδελφοι και συνάδελφοι που ήταν υπέρ της παραμονής έλεγαν μην παρανεύετε στη συζήτηση και μου φάνηκε τότε σαν να είχε προαποφασιστεί το διαζύγιο. Αλλά ήταν αλήθεια ότι ελάχιστες θεσμικές φωνές από την Ευρώπη έλαβαν μέρος στην εκστρατεία πριν το δημοψήφισμα. Τώρα τι γίνεται, είμαστε πιο πιστικοί μετά το δημοψήφισμα, δεν ξέρω, εγώ αμφιβάλλω. Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος πάντως και βέβαια αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εξάλλου δεν έχουμε και πολλές ε, ευκαιρίες και κάποιοι συνάδελφοι ήδη έχουν φύγει από τους Βρετανούς συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήταν υπέρ της παραμονής. Οι συνάδελφοι ακόμα και από τους εργατικούς παρόλο που ήταν ε, υπέρ της παραμονής έφυγαν. Πάντως και αν κάνουμε έτσι είναι τα πράγματα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών είναι να ακούσουμε τι ανησυχίες των συμπολιτών μας, να προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι μια πολιτική υφή σε αυτές τις ανησυχίες ώψη των διαπραγματεύσεων που επιτέλους ξεκίνησαν. Επιτέλους ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε, αλλά τέλος πάντων Ίσως να μου διαφεύγει κάτι, αλλά δεν καταλάβα γιατί χρειάστηκε ένας χρόνος να ξεκινήσει αυτή η δικασία, αλλά εντάξει, εξαρτάται του Βρετανούς πάντα, όχι από εμά. Α, τέλος πάντων. Ένα χρόνο ολόκληρο λοιπόν προσμέναμε το αποτέλεσμα αυτή τη συζήτηση. Τι γίνεται, επαναλαμβάνουμε το δημοψήφισμα, ξεκινάμε διαπραγματεύσει. Δεν ξέραμε. Τέλο πάντων, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το να δώσουμε μια πολιτική μορφή στι ανησυχίε που εκφράζουν οι Βρετανοί πολίτες που ζουν σε άλλες ε, χώρες, μέλη, από τους Ευρωπαίους επίσης που ζουν στη Βρετανία, για να εισακουστούν όλα αυτά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το θεματολόγιο παρουσίασε ο διαπραγματεύτη μας, ο κ. Μπαρνιέ, είναι ξεκάθαρο. Προτεραιότητα θα δοθεί στα δικαιώματα και για τους Βρετανούς που ζουν στην Ευρώπη, αλλά και για τους συμπολίτε μας Ευρωπαίους που θέλουν να συνεχίσουν να διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία και όπως είπαμε το πρωί ίσως θα έχουμε ένα, πολύ πιθανώς να έχουμε ένα ψήφισμα δικό μας το οποίο θα επικεντρωθεί σε όλες αυτές τις ανησυχίες που αφορούν το καθεστώς των Ευρωπαίων στη Βρετανία, που είναι πολλοί και ανησυχούν και βεβαίως είμαι υπέρ το να διατηρήσουμε ανοιχτές αυτές τις αναφορές και να τους δώσουμε μια πολιτική μορφή, η δομή. Γιατί πραγματικά οι Ευρωπαίοι πολίτε θεωρούν ότι είναι δική μας ευθύνη όταν μας γράφουν. Η κυρία Μπεθέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω την αναφέρουσα για την συγκινητική της παρέμβαση. Ήταν υποδειγματική. Όταν έρχονται οι αναφέροντες εδώ στην Επιτροπή μας, μας εμπνέουν και μας ενισχύουν, μας δυναμώνουν στη σχέση μας, την αμοιβαία. Είμαστε το ανοιχτό παράθυρο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και οι Βρετανοί πολίτες και οι Ευρωπαίοι πολίτες που είναι στη Βρετανία Έτσι μας βλέπουν ακόμα και τουλάχιστον για δύο χρόνια. Να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, κανόνες του παιχνιδιού δεν μπορούν να αλλάξουν. Καθοδόν. Και σε σχέση με αυτά που είπε ότι είναι ένα θέμα εμπιστοσύνης. Οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο λιγότερο τους ερετούς, τα κοινοβούλια, την εκκληστική εξουσία. Και νομίζω ότι οι Βρετανοί που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχασαν την εμπιστοσύνη τους, ιδιαίτερα μετά τα αποτελέσματα που είδαμε στις πρόσφατες εκλογές. Και με την κακομεταχείριση και έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται να έχασαν την ε, δυνατότητα να αποτελούν ακόμα μια απειλή αυτή η αιρετή των Βρετανών. Πάντως φαίνεται ότι θα ζητηθεί από τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία να καταγραφούν. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται όσο έχουμε συγκεκριμένου κανόνες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν χρειαζόταν να καταγραφούν. Γιατί απλούστατα σου είχαν πει δεν χρειαζόταν. Οποιαδήποτε λοιπόν πρωτοβουλία υιοθετήσει μονομερό η Βρετανική κυβέρνηση όσο διεξάγονται οι διαπραγματεύσει δεν έχει καμία ισχύ. Και καταλήγοντα. για να μην μακρηγορώ, επειδή θέλουμε να δώσουμε εδώ στην Επιτροπή το λόγο στους πολίτες, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισάκουσε τις ανησυχίες, αλλά πέραν αυτό που έλεγε ο συνάδελφο Μπρέντα, θεωρώ ότι είμαστε ένα χώρο όχι μόνο συζήτηση, τοποθέτηση και λήψη πολιτική θέση. Είμαστε ένα νομοθετικό κοινοβούλιο, το οποίο συνομοθετεί μαζί με το Συμβούλιο, αλλά νομοθετεί και είμαστε ιερετοί. Ιερετοί εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Οπότε αυτή η Επιτροπή και άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από κοινού έχουμε καθορίσει ακριβώς το πλαίσιο δράσης και για πρώτη φορά πετύχαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη με όλα τα θεσμικά τη όργανα εθαγραμμίζεται με ένα κοινό στόχο. ότι το πρώτο, οι πολίτε δεν είναι ένα σλόγγαν απλό και μόνο, είναι μια δήλωση αρχή Οι αρχών. Και οι πολίτε, όπως λέγαμε το πρωί, έχουν μετατραπεί σε κάτι το απτό, δηλαδή ε, με μια μορφή και μια ιστορία μετά το Brexit. Το έτος ένα λοιπόν του Brexit βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Οπότε θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ανυποχώρητοι και να μετατρέψουμε αυτό το πρώτο επολίτε σε κάτι το απτό και σε κάτι που αποτελεί μια εγγύηση δικαιωμάτων. Αλλά επιπλέον, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, να πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι αυτή η απόφαση που λήφθηκε υπό τις συνθήκες που γνωρίζουμε όλοι είναι ανατρέψιμη, ότι μπορούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα. Υπάρχει δυνατότητα και νομική και πρακτική, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να σκεφτεί τους πολίτες και το μέλλον του στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που είναι ένα έτος αργότερα. Είναι νέο. Το καλό των πολιτών είναι αυτό που υπερέχει και αν εμείς δεν κάνουμε την δουλειά μας, δηλαδή να λύνουμε τα προβλήματα, τότε είμαστε άχρηστοι. Οπότε ευχαριστώ τους εκατοντάδες πολίτες που εκπροσωπούν πολλούς άλλους περισσότερους που κατέβαλαν αυτές, κα, ε, κατέθεσαν αυτές τις αναφορές. Θεωρώ ότι θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση σωστά και να δώσουμε σωστές λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το σημείο λέγοντα πω η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή, θα παρακολουθούμε τι διαπραγματεύσει και μόλις έχουμε κάποια συγκεκριμένα ε, στοιχεία τότε θα σας καλέσουμε ξανά και θα συνεχίσουμε την πορεία της αναφοράς. Η αναφορά λοιπόν θα μείνει ανοιχτή μέχρι να υπάρξει κάποια συμφωνία ανάμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Αναφορά 101-2017 του Τόνι Venables, Βρετανικής Ιθαγένειας και πάλι αφορά το Brexit. Από όσο γνωρίζω, ο αναφέρον είναι εδώ. Κύριε Βένεμπολς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι μαζί με τον Ρότζερ Κασάλε, ο οποίος είναι ο ιδρυτής των New Europeans και είναι πολύ δραστήριος, προσπαθεί να ε, δημιουργήσει ένα μεγάλο λόμπι που να ασκήσει πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι... Νομίζω πως και άλλοι αναφέρονται στο είπαν. Εμείς θεωρούμε πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο ένα διάβλος ε, και ένα βήμα όπου μπορούμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας ε, για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η αναφορά μου έχει ως θέμα, μάλλον έχει ως σκεπτικό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο, είναι το μόνο ε, εκλεγμένο θεσμικό όργανο και γι' αυτό μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει θέση για το θέμα της ε, υπηκότητας και είναι τόσο σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, όχι μόνο ως ε, φύλακα των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και ε, ως φύλακας της ασφάλειας γενικότερα. Οι συνθήκες αναφέρουν ότι όποιο άτομο έχει ε, την επικότητα ενός κράτους μέλους Ένωσης είναι πολίτης της Ένωσης. Όμως οι συνθήκες δεν λένε πώς γίνεσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής, ε, μάλλον αναφέρουν πώς γίνεσαι πολίτης, ε, όμως δεν αναφέρουν τίποτα για το τι συμβαίνει αν χάσεις την ε, υπηκότητα της Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ποτέ δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί, είναι πάντα αφορμή για διαξυφισμούς, έντονες συζητήσεις, τα κοινοβούλια, είναι τροφή για τα συνταγματικά δικαστήρια. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ακολουθήσει αυτή την πορεία. Να πω επίσης ότι κανείς δεν πρέπει να στερηθεί την υπηκότητά του και χωρίς, χωρίς κάποιον κοινοβουλευτικό έλεγχο προηγουμένως, χωρίς να ενημερωθεί εκ των προτέρων, χωρίς να έχει το δικαίωμα έφεσης, χωρίς να του δοθούν εναλλακτικές λύσεις. Και δεν υπάρχει άλλο θεσμικό όργανο ε, πέραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορεί να ασχοληθεί με το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Γιατί λοιπόν παραμένει άλλη το, το θέμα, για τρεις λόγους. Πρώτα, εάν η πλειοψηφία των Βρετανών είχε ψηφίσει να απαρνηθεί την ευρωπαϊκή της ηθαγένεια, θα βρίσκαμε κάποιες ενδείξεις, θα τις βλέπαμε πριν το δημοψήφισμα. Ένα, η επιστολή που έστειλε η Βρετανική κυβέρνηση σε κάθε νοικοκυριό, αν την διαβάσετε, αν διαβάσετε όλες τις ε, πληροφορίες που, και τους κανόνες ε, τον, πριν το δημοψήφισμα, δεν θα βρείτε απολύτω τίποτα για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Μόνο τώρα προέκυψε το θέμα αυτό. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το πρώτο δικαίωμα, η ελεύθερη κυκλοφορία δηλαδή των πολιτών ε, εντό ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ στην ε, εκστρατεία πριν το δημοψήφισμα. Τώρα το να αμφισβητήσεις ένα δημοψήφισμα δεν είναι τίποτα άλλο ε, παρά να ίσω με το να πεις ότι λείπουν στοιχεία. Δεν μας είπαν όλη την αλήθεια. Έπειτα, εκείνοι που επλήγησαν πολύ, ε, περισσότερο από όλους δεν είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν, να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα. Εγώ ζω στο εξωτερικό πάνω από 15 χρόνια, δεν έχω το δικαίωμα να ψηφίσω στη χώρα μου. Και αυτό δεν είναι ψηλό πράγματα. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια μπορεί να αλλάξει ζωές. Ε, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μου. Έχω χτίσει την προσωπική και επαγγελματική μου ζωή βασισμένο σε αυτό, ε, τη δουλειά μου. Μέχρι και την ε, πνευματική μου ζωή, αν θέλετε. Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, μπορώ να σας στείλω βιβλίο να διαβάσετε για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Τώρα, είναι φυσιολογικό να στερείται κάποιο την ηθαγένειά του όταν δεν έχει καν το δικαίωμα να ψηφίσει γι' αυτό και να αποφασίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάποιοι θα πούν ότι δεν ήταν και η καλύτερη διαδικασία, η δημοκρατία έτσι και αλλιώς δεν είναι τέλεια, όμως έχει καμιά σημασία. Έχει έχει διότι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν είναι μια μαριονέτα στα χέρια εκείνων που παίρνουν αποφάσεις. Και μάλιστα η μαριονέτα πάπε on a String ήταν ένα τραγούδι με το οποίο κερδίσαμε τη Eurovision κάποτε. Αλλά να αναφερθώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πω πόσο έλαμψε δια της απουσίας του μέχρι τώρα. Διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περιπτώσεις όπως η αντίον ε, η περίπτωση υπόθεση Σαμπράνο ε, έχει βασική λειτουργία, θεμελιώδη λειτουργία. Το έχει αποδείξει αυτό. Αυτές οι περιπτώσεις ήταν οι πρώτες περιπτώσεις ε, διεθνούς, διεθνικής ηθαγένειας. Και τώρα, ολοένα και περισσότεροι, κυρίως νέοι, έχουν άμεσες επιπτώσεις από τις συνέπειες του ε, δημοψηφίσματος, της αποχώρησης. Το ευρωπαϊκό όνειρο φθήνει. Τέλος, νομίζω πως αυτή η αναφορά είναι πάρα πολύ σημαντική και για δύο λόγους. Αμέσως μετά το δημοψήφισμα, αντέδρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκανε μια πρόταση για ε, μια διαφορετική μορφή ηθαγένειας, μια έτσι, συνδεδεμένη μορφή ηθαγένειας. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. αλλά πρέπει να κάνετε μία επιλογή. Το είπε και η Ντανούτα Χούμπνερ νωρίτερα. Μπορείς να διατηρήσεις όλα αυτά τα δικαιώματα που έχει ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που ακούμε εδώ και αυτά που ανέφερε η Τερίζα Μέη ή προσπαθεί να πάρει. Μπορείς λοιπόν να τα κρατήσεις χάνοντας την ιδιότητα του μέλους. Ε, μπορώ να σας πω από την επαγγελματική μου εμπειρία ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μία γενιά ανθρώπων οι οποίοι στο μέλλον θα έχουν τρομερά προβλήματα. Δεν θα μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους, δεν θα μπορούμε να ενημερώσουμε, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και διοικητικά ε, και άλλου τύπου. Δεν έχουμε τους πόρους αυτή τη στιγμή να χειριστούμε αυτά τα 5 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε όλη την επικράτεια της Ένωσης σε διαφορετικό κράτος ε, από εκείνο το οποίο προέρχονται. Και μας είπατε για θεμελιώδη βασικά δικαιώματα. Αυτά. Υπάρχουν και άλλα. Ακούσαμε και την μελέτη σήμερα το πρωί. Υπάρχουν όλες αυτές οι απρόβλεπτες ε, περιπτώσεις, υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες του καθενός ε, που τον καθεστούν μοναδικό στην προσωπική, την επαγγελματική του ζωή. Νομίζω πως εδώ δημιουργούμε μία γενιά δυσαρεστημένων. Απ' την άλλη, εάν ακολουθήσουμε αυτό που ανέφερε διακριτικά η Ντανούτα Χούμπνερ, δηλαδή αυτά περί ευρωπαϊκής ηθαγένειας, αν μπορούσαν να κρατήσουν οι πολίτες αυτοί το καθεστώς του Ευρωπαίου πολίτη, τότε αντί να τσακωνόμαστε για δικαιώματα, για λεπτομέρειες, θα έχουμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε το ε, καθεστώς μας. Και αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, το δικαστήριο, είναι θέματα ηθαγένειας. Υπάρχει και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βασικά δικαιώματα, όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί. Εξαιρετικό είναι το κείμενο αυτό, δεν αναφέρει όμως καθόλου την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και εάν υπάρχει ένα θεσμικό όργανο που θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους αν έχουν ερωτήσεις ή να πούν κάτι κύριε Γιάρ. Επειδή το θέμα ε, διατρέχει όλη τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να είναι όπλο στην διαπραγμάτευση. Όταν μιλάμε για μια ευρωπαϊκή υπηκότητα δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο Brexit γιατί κάποιοι ε, και εγώ ε, μεταξύ αυτών ε, θεωρήσαμε ότι δεν θα υπάρξει Brexit. Οπότε δεν μας απασχόλησε το θέμα γιατί λέγαμε δεν θα γίνει Brexit. Και οι άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονταν για το Brexit δεν το θεωρούσαν θέμα. Γιατί δεν είναι και ωραίο θέμα αν θέλει κανείς το Brexit. Εγώ ανήκω σε αυτούς που λένε ότι θα πρέπει να προσέξουμε τα δικαιώματα των πολιτών και στις δύο πλευρές να γίνουν σεβαστά οι πολίτες ε, της ε, Μεγάλης Βρετανίας που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστρόφως. Οπότε η ιδέα αυτή τη συνδεδεμένη υπηκότητα δεν έχει φύγει. Αλλά βεβαίως ε, πρέπει να το δούμε ως ένα πακέτο. Ο είπε πριν ότι δεν επιτρέπεται να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αρκετά πράγματα να διαπραγματευτούμε, οικονομικά κτλ. Αλλά όχι κάτι άλλο. Και βεβαίω δεν θα ωφελήσει καθόλου και το αποτέλεσμα. Οπότε πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Δηλαδή θα πρέπει να διατηρήσουμε τα δικαιώματα τα οποία δημιουργήθηκαν ε, και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τα θέσουμε και στην Βρετανική κυβέρνηση και στους δικούς μας τους διαπραγματευτές, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να μην ε, το παραβλέψουμε. Σας ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ κυρία συνάδελφα μια πρακτική πρόταση. Ξέρω πως εκτός από αυτήν την αναφορά υπήρχε και ένα έγγραφο που ανέφερε τα ζητήματα αυτά και τα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα μπορούσαμε νομίζω να το αποστείλουμε και σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το ψήφισμα αυτό. Έτσι θα μπορέσει ακριβώ ε, η αναφορά αυτή να παίξει ρόλο στην διαδικασία. Ναι. Συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι. Να πω λίγο κάτι για το θέμα της ε, δημοκρατίας. Ε, είναι κάτι το σημαντικό το οποίο έχει συζητηθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι το έχουμε πλήρως αντιληφθεί. Γιατί οι πολίτες του Ηνωμένου Βασίλειου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Το δικαίωμα ψήφου αφορούσε μόνο τους Βρετανούς πολίτες. Αυτά τα 3,5 εκατομμύρια λοιπόν άτομα τα οποία κατοικούν και κατοικούσαν και πολύ καιρό ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν για το μέλλον τους κάτι το οποίο είναι ε, πραγματικά παράδεκτο και πολύ διαμαρτυρηθήκαμε τότε νομίζω λοιπόν πως όταν θα συντάξουμε το ψήφισμα πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά γιατί οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά στερήθηκαν αυτό το δικαίωμα Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Σας ευχαριστώ κύριε Venables. Θα παρακολουθήσουμε την ε, κατάσταση και θα σας ε, ενημερώσουμε. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου κάθε αναφορά καταγράφεται στα πρακτικά και θα διαβιβαστούν όλα αυτά στον κύριο Μπαρνιέ. Γι' αυτό είναι σημαντικά όλα αυτά. Γιατί θα διαβιβαστούν και στην ε, Κομισιόν και θα παρακολουθήσουμε τα πράγματα πολύ προσεκτικά. Γι' αυτό ακριβώς ε, πρέπει να είμαστε σήμερα πολύ προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Βέναμπλς και θα συνεχίσουμε τον διάλογο όταν έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ρόμπερτ. Ναι. Ρόμπερτ Βέστερνι. 08 δεν βρίσκεται εδώ αναφέρον. Ο συνάδελφος Κόρμπιτ τον εκπροσωπεί. Ευχαριστώ. Κύριος Western ζητά συγγνώμη. Θα έχετε δει πως αναφέρον λέει ότι αυτός και πολλοί άλλοι αν γίνει το Brexit θα στερηθούν ε, την ευρωπαϊκή τους υπηκότητα παρά τη θέλησή τους. Ε, κάτι ε, βεβαίω ακόμη πιο φρικτό για όσους ψήφισαν να παραμείνουν ή όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Αναφέρω λοιπόν κάνει μια παρομοίωση με την εθνικότητα και ξέρει ότι δεν είναι το ίδιο, αλλά λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο, τα άρθρα 15 και 17 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λέει εκεί ότι κανείς δεν θα στερηθεί αυθαίρετα την υπηκότητα του. Υπάρχουν κάποιες εγγύησεις ε, για τους ε, πολίτες. Και λέει Κατά αναλογία, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ζητάει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο να επιτρέψει στους Βρετανούς πολίτες που θα το ζητήσουν να διατηρήσουν την Ιθαγένεια μετά τον Brexit, αν λάβει αυτό χώρα. Λοιπόν, βλέπω ότι η πρόταση που έχουμε τώρα διαδικαστικά είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να την στείλουμε σε μια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Συνταγματικών Υποθέσεων και αυτό είναι το σωστό. Εάν απαιτείται αλλαγή της συνθήκης, τότε πράγματι η Επιτροπή Συνταγματικών είναι η αρμόδια. Αλλά εάν είναι δυνατόν, όπως μας είπε ο κύριος Βέναμπλς να παραμείνει αυτή η δυνατότητα χωρίς αλλαγή της συνθήκης τότε πρέπει να το δει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πρέπει να εξετάσουμε και τις δύο δυνατότητες εν πάση περιπτώσει ο κύριος Φερχόφστα τόσο εκπρόσωπός μας στην διαδικασία του Brexit θα ενημερωθεί όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, ήδη έχει εκφράσει μεγάλο ενδιαφέρον. για τις ε, δυνατότητες αυτές. Να πω πως όλες αυτές οι αναφορές ε, δείχνουν μια βαθύτατη ανησυχία μεταξύ πολλών πολιτών ε, που ζουν είτε στην Ένωση είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο αισθάνονται Ευρωπαίοι, θέλουν να κρατήσουν αυτή την σύνδεση. Αυτό είναι θέμα βεβαίω και συναισθηματικό, αλλά και θέμα λογική. Υπάρχουν κάποια νομικά δικαιώματα τα οποία βεβαίω θα χαθούν εάν γίνει το Brexit. Που είναι θέμα τη ευρύτερη συζήτηση των δικαιωμάτων των πολιτών. Ο μόνο τρόπο για να είμαστε σίγουροι ότι θα διατηρήσουμε όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα είναι να σταματήσει το Brexit. Υπάρχουν άτομα στην Βρετανία βεβαίως που υποστηρίζουν κάτι τέτοια και θα ήθελα να σα παρακαλέσω να ενταχθείτε στο ευρωπαϊκό κίνημα της Βρετανίας που βεβαίω προσπαθεί να σταματήσει το Brexit μαζί με άλλε οργανώσει, αλλά αν δεν συμβεί αυτό εάν συμφωνήσουμε για το Brexit σε λιγότερο από δύο χρόνια σήμερα, θα έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου για έγκριση ή απόρριψη. Και το Κοινοβουλίο, το οποίο έχουν εκλέξει οι πολίτες, βεβαίως ε, θα θεωρήσει ότι θα πρέπει να κοιτάξει ειδικά το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών και στις δύο περιπτώσεις. Και ε, πρέπει να θυμόμαστε κάτι. Πέρα από το ναι ή όχι, το Κοινοβούλιο έχει την επιλογή, όπως και οποιαδήποτε εθνική κυβέρνηση, να αναπέμψει την συμφωνία στο δικαστήριο και να ζητήσει από το δικαστήριο εάν αυτή η συμφωνία είναι σύμφωνη με τις συνθήκες και την χάρτα δικαιωμάτων. Και ε, μετά βεβαίω έχουμε το άρθρο 15. Έχουμε λοιπόν την συμφωνία αυτή που θα υπάγεται στο άρθρο 50, που είναι θέμα άρα κοινοτικού δικαίου. Πρέπει να σέβεται την χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία από αυτό, το κοινοβουλίο θα πρέπει να είναι έτοιμο να αναπέμψει την συμφωνία στο δικαστήριο πριν ψηφίσει ναι ή όχι ομολογουμένως θα χρειαστεί λίγος χρόνος, το δικαστήριο θα πρέπει να πει ότι σταματάει τώρα το χρονόμετρο, αλλά αυτό είναι διαδικαστικό. Αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι πολύ πιο ουσιαστικό, είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Για μένα και off the record, έτσι. Αυτή η αναφορά μπορεί να γίνει αφορμή να μιλήσουμε για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Πολιτικά όμως είναι πολύ επικίνδυνο πιστεύω εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σταματήσει, βάλει ένα φρένο σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν. Ε, όσοι υποστηρίζουν το Brexit θα πούν ότι μας αναγκάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε. Μας πιέζουν. Αλλά ας περιμένουμε μέχρι το 2019 που θα έχουμε κάτι χειροπιαστό, θα έχουμε μια συνθήκη, να δούμε μετά τι θα σημαίνει αυτό, αυτή η αποχώρηση για τους Βρετανούς. Αλλά δεν μπορεί να, μια οργάνωση πολιτών να πάει στη Βρετανική κυβέρνηση και να πει όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό, δεν συμφωνούμε, θέλουμε δημοψήφισμα και μετά το 2019 να γίνει άλλο δημοψήφισμα που να πει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο όχι άλλαξε γνώμη, θέλει να παραμείνει. Όπως ε, είπα και πριν, μόνο οι Βρετανοί μπορούν να αλλάξουν αυτή την απόφαση. Αυτό είναι ο μόνος δρόμος, αλλά αυτή είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Φυσικά πιστεύω πως δεν έχει λήξει ακόμα το θέμα. Αυτό το δημοψήφισμα πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, όμως στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο ε, δεν νομίζω πως ε, μπορούμε ή έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε αυτή την διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και θα δώσω το λόγο σε, σε Ναι, δεν σας πειράζει να απαντήσω σε αυτό που είπατε. Βεβαίως πολιτικά θα ήταν καλό να ή καλύτερο να σταματήσει το Brexit, αλλά αυτό μόνο από τη Βρετανία μπορεί να προέλθει αρχικά. Αλλά αυτό που είπα για το να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το Brexit θα πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών και από τις δύο μεριές, και των Βρετανών και αυτών της Ευρώπης που διαμένουν στη Βρετανία γιατί και τα δυο τα δικαιώματα μπορούν να επηρεαστούν από αυτή τη συμφωνία. Ανεξάρτητα λοιπόν από το τι θα συμβεί, κατά πόσο θα σταματήσει ή όχι η διαδικασία του Brexit, ανεξάρτητα από αυτό τέλο πάντων, εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε το ότι δεν θα χάσουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Είμαστε μια επιτροπή που έρχεται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να συζητούμε το θέμα, το βάζουμε στη μίληση διάταξη συνεχώ. παραμένει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά και θα επανέλθουμε μόλις ε, έχουμε περισσότερα, περισσότερες Επόμενη αναφορά... Από τον Edward Williamson. Επίσης, για το Brexit, ο Νοφέρον είναι εδώ και του δίνω αμέσω το λόγο. Sorry, ε, is Mr. Williamson here? Yes. Δεν είναι εδώ ο κύριος Williamson, αλλά εδώ είστε. Ναι, ναι, ωραία. Έχετε το λόγο. Μ' ακούτε? Ωραία, ευχαριστώ. Υποβλήθηκε αυτή η αναφορά το Σαββατοκύριακο μετά το δημοψήφισμα. Έχουν καλυφθεί φαντάζομαι αρκετά θέματα, αλλά τόσο πάντων θα σα παρουσιάσω ακριβώ το σκεπτικό. Λάβαμε υπόψη λοιπόν τις διάφορες ε, επιπτώσεις αυτής της πολιτικής πράξης που ανοίγησε μετά το referendum και τι επιπτώσει τη. Δεν θα ε, επισέλθω στις επιπτώσει όσον αφορά τη συνθήκη. Είμαι εδώ απλά και μόνο να παρουσιάσω, για να παρουσιάσω το δικό μου το αίτημα. Σήμερα το πρωί ακούσαμε από διάφορους πολίτες Βρετανούς που ζουν στην Ένωση τις απόψεις τους και αντίστροφα πολίτες της Ευρώπης που μένουν στην Βρετανία κάποια πράγματα για τις επιπτώσεις του Brexit. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό επίσης να ακούσουμε και τους Βρετανούς που ζουν στη Βρετανία και που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να υλοποιήσουν, να εφαρμόσουν τις αρχές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. ανεξάρτητα από το τι αποφασίζουν να κάνουν οι κυβερνήσεις. Επίσης, να πω ότι το κίνητρό μου δεν είναι πολιτικό. Σήμερα είδα ότι ακούσαμε πολιτικές τοποθετήσει από τους εργατικούς, από το Συνφρέιν νωρίτερα που έκαναν τοποθετήσει. Αυτή η συζήτηση ίσως να δημιούργησε κάποιες δικοφιλίες, αλλά τουλάχιστον μεταξύ των δικών μου γνωστών του κύκλου μου, αν είναι καλό ανέκυψε, είναι ότι συζητήθηκε παντού αυτό το θέμα και διαφορετικά, αλλά είχαν προκύψει όλα αυτά, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι εψαχόμαστε σε μια φάση εμφαλοσκόπησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και ελπίζω κατά διάρκεια αυτής της περίοδου να αποκαταστήσουμε τη λογική και τις δημοκρατικές παραδόσεις στη χώρα μου. Πάντως, οποιαδήποτε θέση της Ένωσης εφαρμοστεί για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια είτε στη Βρετανία είτε στην Ένωση ελπίζω να επουλώσει τις πληγές αυτής της πολύ διχαστικής διαδικασίας. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι γενναιόδωρο και μεγαλόψυχο ενώπιον προκλήσεων μικροπρεπών. Αυτό μπορεί να φαίνεται προφανές ή εύλογο, αλλά δεν ξέρω πόσοι από διαβάζουν τον, τον τύπο, τον καθημερινό, το, το tabloid στην Αγγλία. Θα δείτε ότι δεν είναι το μοναδικό θέμα πολιτικής συζήτησης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Βρετανία, συγγνώμη. Επίσης, Αναρωτιέμαι κατά πόσο οι πιθανέ πολιτικέ λύσει στη Βόρεια Ιρλανδία σε σχέση με την Συμφωνία τη Παρασκευή. Αν λοιπόν οι λύσει για του πολίτε τη Βόρεια Ιρλανδία αναρωτιέμαι κατά πόσο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στου πολίτε τη Βρετανία ή συνολικότερα του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι καταλαβαίνω, η συζήτηση για τη Βόρεια Ιρλανδία είναι βέβαια κάπως εξειδικευμένη αλλά νομίζω ότι ίσως να χρειαστεί να τετραγωνίσουν τον κύκλο και ελπίζοντα, ελπίζω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας να προκύψουν κάποια διδάγματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στους υπόλοιπους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τους ευρωβουλευτές μας της Βρετανίας να είναι περισσότερο παρόντες και να συμβάλλουν στην ανέβρεση συμφωνίας. Ξέρω ότι να συζητήσει τον Ομέρο Βασίλειο διακομματικά για αυτό το θέμα. Αλλά πιστεύω ότι το θέμα αυτό ξεπερνάει τα μικροκομματικά, αφορά αρχές και αξίες και φαίνεται ότι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κομμάτι της συζήτησης ακόμα ακολουθεί μικροκομματικές σκοπιμο, σκοπιμότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα ζητούσα από τους εκπροσώπους που είναι εδώ του, Βρετανικού Κοινοβουλίου να συμβάλλουν και να προσπαθήσουν να πείσουν τους ομολόγους τους, τους συναδέλφους τους. Ίσως επίσης είναι καλό να ακούμε βέβαια και αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη και το πρόβλημα είναι ότι καμιά φορά εδώ πέρα εδώ στη συζήτηση αυτή έχω την εντύπωση ότι μιλάω στους μοιημένους και ίσως να αμφιβάλλει κανείς την χρησιμότητα αυτών των συζητήσεων. Να πω, καταλήγοντας, ότι υπάρχουν διάφορα θεσμικά περίπλοκα ζητήματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί αλλά βεβαίως θα πρέπει να περιλάβουμε όλους τους Βρετανούς πολίτες σε οποιαδήποτε συμφωνία συναυθεί μελλοντικά. Είτε ακολουθήσει την πεπατημένη συμφωνία, συμφωνησιακής ή οποιαδήποτε άλλη λύση. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε ανυποχώρητοι σε αυτό και να μην ε, τους προσεγγίσετε αυτούς τους πολίτες ως απλά και μόνο διαπραγματευτικό χαρτί. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ακούω αυτά που λέτε. Προσέχω και βλέπω πως πολύ συχνά, κάθε δύο εβδομάδες, μια φορά το μήνα, γίνεται μία ακρόαση με θέμα το Brexit. Πάντα το Κοινοβούλιο προσέχει και παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, ε, ρωτά να μάθει την παραμικρή λεπτομέρεια. Ένας φίλος μου είναι νομικός, ειδικεύεται στο διεθνές δίκαιο και μου είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ε, ανοιχτά θέματα, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία που ε, μπορεί να διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, δεκαετίες ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι εύκολη σε καμία περίπτωση. Και οι Βρετανοί πολίτες μπορεί στο τέλος να συνειδητοποιήσουν ότι έκαναν λάθος. Και θα ήθελα να πω στον αναφέροντα ότι καλύτερα να αλλάξεις μία άσχημη άποψη. Γι' αυτό δεν πρέπει να απογοητεύεστε. Είναι στο χέρι του Βρετανικού λαού, αλλά θα δώσω τώρα το λόγο στην συνάδελφο που τον ζήτησε. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Βίλιαμσον, ο οποίος μάλιστα είναι και από τη δική μου εκλογική περιφέρεια, το Λονδίνο. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια για το Λονδίνο και τις άλλες μεγάλες πόλεις το Ηνωμένου που ψήφισαν να παραμείνουμε στην Ένωση. Το Λονδίνο ψήφισε να παραμείνει με 60%. Η Σκοτία ψήφισε να παραμείνει στην Ένωση. Ο κύριος Βουίλαμσον μας είπε για ε, διχασμό του Βρετανικού λαού. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό, παρότι είναι λίγο εκτός θέματος. Υπάρχει λοιπόν ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε ύπεθρο και αστικά κέντρα, σε και σε βιομηχανικά, ή πρώην βιομηχανικά κέντρα. Υπάρχει μία σαφή στάση για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως ε, αυτή η Επιτροπή ίσως ε, θα ήθελα να μάθει ότι υπήρχαν διάφορες δημοσκοπήσεις, έγιναν πρόσφατα, που έδειξαν ότι η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει ε, άποψη για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι τώρα μετανιώνουν την απόφαση να αποχωρήσουν. Κινούνται λοιπόν τα πράγματα και νομίζω πως αυτό είναι ζωτική σημασία για τη δημοκρατική διαδικασία. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο ένα φωτογραφικό αποτύπωμα μια στιγμή είναι κάτι που συνεχώς μεταβάλλεται, αλλάζει και πρέπει να καταλάβουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Ε, κατά μία έννοια έχετε δίκιο. Οι Βρετανοί είναι αυτοί που μπορούν να πάρουν την οριστική απόφαση, όμως ε, αποχωρούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ε, τουλάχιστον την δυνατότητα να τοποθετηθεί, να έχει ίσο δικαίωμα με τους Βρετανούς. Εάν εσείς ε, θεωρείτε ότι το δημοψήφισμα ήταν απόλυτα δημοκρατικό, τότε επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Αυτή η απόφαση πάντως έχει διχάσει ε, τον κόσμο και όλο ένα και περισσότεροι Βρετανοί έχουν μετανιώσει την απόφαση που ελήφθη. Και τα πράγματα φυσικά δεν ε, βελτιώνονται με μια κυβέρνηση μειοψηφία η οποία σκοπεύει να παραμείνει στην αρχική της γραμμή και ο κύριος Βίλαμσον αναφέρθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει γιατί η υπόλοιπη Ιρλανδία παραμένει μέλος της Ένωσης. Πρέπει να λυθεί λοιπόν το θέμα για να παραμείνουν τα σύνορα ανοιχτά στην Ιρλανδία. Είναι μία από τις πολλές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε και τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα ε, τώρα με την κατάρρευση της ε, συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Υπάρχει λοιπόν ε, πολύ μεγάλη βαρύτητα στις αποφάσεις που λαμβάνονται και το δημοψήφισμα εγώ προσωπικά πιστεύω πως ε, δεν είναι οριστικό και αμετάκλητο και χρειάστηκε Χρειάστηκαν 40 χρόνια για να φτάσουμε ως εδώ. Νομίζετε πως θα τόσο εύκολο να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι που μαζεύτηκε σε 40 χρόνια. Είπε και ο κύριος Βίλιαμσον εξάλλου ότι ίσως να μην είναι απόλυτα σχετικό για αυτή την επιτροπή, όμως εγώ θεώρησα πως έπρεπε να τα αναφέρω αυτά γιατί μας αφορά άμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία, όπως και με όλες τις επιτροπές. Εάν κάποια άλλη επιτροπή θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, φυσικά και θα τη στείλουμε την αναφορά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γουίλιαμσον που υπέβαλε αυτή την αναφορά και ειδικά να ευχαριστήσω τους ε, πολλούς ε, Βρετανούς ε, πολίτες που έγραψαν επιστολές σε ευρωβουλευτές, όχι μόνο Βρετανούς ευρωβουλευτές. Και ο Γκίφερ Χόφστατ είπε ότι είχε λάβει εκατοντάδες email από κόσμο που έλεγε ότι δεν ήθελε να χάσει τα δικαιώματα που του έδινε η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και δεν είναι θέμα του ότι ζουν στο εξωτερικό και αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στη ζωή τους, αλλά αισθανόταν Ευρωπαίοι και εκτιμούσαν ακριβώς ε, το ότι υπάρχει κάποια προσθεμένη αξία. Και ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο εστάλει στο Κοινοβούλιο και άλλαξε η ατμόσφαιρα της ε, συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να το ξέρετε αυτό. γιατί η συζήτηση αυτή έγινε μια ευρύτερη συζήτηση όχι μόνο για τα 4,5 εκατομμύρια αυτούς τους ανθρώπους, το 1,5 εκατομμύριο Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν στη Βρετανία. Αλλά έγινε και θέμα του πώς αντιλαμβάνονται οι Βρετανοί αυτούς και πραγματικά συνέβαλε σε μια σημαντική συζήτηση και όταν κάναμε μια ακρόαση πριν από λίγες εβδομάδες ε, για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια από κοινού οι Επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών και Αναφορών ε, προέκυψε σαφώς από την συζήτηση με τον Αγγί Φερχοφθατ η ακρόαση αυτή ήταν ότι είχαμε ε, συμμετοχή από το UKIP και τους ευρωσκεπτικιστές ε, και μας είπαν την άποψή τους για τα ζητήματα αυτά. Και αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι έχουμε πολίτες που έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μιλάνε με ευρωβουλευτές ευρωβουλευτές που έλεγαν να φύγουμε από την Ένωση και δεν έχουν τον χρόνο, το θάρρος να μιλήσουν ε, πρόσωπον πρόσωπο με τους πολίτες αυτούς. Αυτό θεωρώ ότι είναι άδικο πραγματικά για ανθρώπους οι οποίοι υποβάλλουν ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάξει, μπορεί να είναι κάπως κομματικό αυτό που λέω, αλλά πρέπει να πούμε ότι εμείς, εσείς αφιερώσατε χρόνο να αρθείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιοι ευρωβουλευτές ε, που αφιέρωσαν χρόνο και χρήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δυσφημίσουν την Ένωση θα μπορούσαν να πούν τουλάχιστον γιατί είναι κατά της ε, Ένωσης. Ναι, με ακριβώς το και θα προετοιμάσουμε ένα ψήφισμα και θα φροντίσουμε στο ψήφισμα αυτό να μην έχουμε μόνο τις ανησυχίες των 4,5 εκατομμυρίων αλλά και των Βρετανών στην Βρετανία που θέλουν ε, να διατηρήσουν ε, την ηθαγένεια και τα δικαιώματα τους γιατί δεν είναι εύκολο συνταγματικό ερώτημα και άνθρωποι όπως ο Ρίτσαρντ που βεβαίως ε, μας συμβουλεύει για αυτά ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι ότι υπάρχουν εκατομμύρια Βρετανών που θεωρούν ότι χάνουν κάτι ακόμα και αν παραμείνουν στη Βρετανία. Πίτερ. Ναι, να συμπληρώσω. Η δική μου η ομάδα, εντάξει δεν έχει καθόλου Βρετανούς, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα ήθελα να αναφέρω ότι όταν είχαμε τους μεγάλους τίτλους που έλεγαν Brexit means Brexit, η δικιά μου ομάδα πάλεψε έτσι ώστε να μπει στο ψήφισμα και η πιθανή αναστολή του, του Brexit. Δηλαδή μπορεί και ένα διαζύγιο ακόμα να ανακληθεί θεωρητικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω και σας και τους αναφέροντες να συνεχίσετε και εδώ και στην χώρα σας γιατί χρειάζεται αυτή η ατμόσφαιρα της συζήτησης. Και... Νομίζω πως όλα τα γεγονότα, τα επιχειρήματα είναι κατά του Brexit, παρόλα αυτά αυτό αποφασίστηκε. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσετε να γνωστοποιείτε τα προβλήματα, όχι μόνο εδώ, εδώ θα σας βοηθήσουμε οπωσδήποτε στις Βρυξέλλες, αλλά και στη Βρετανία, γιατί πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση. Ε, πρέπει να προσέξουμε να μην πληγούν εδώ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Λοιπόν, οι αναφορές είναι σημαντικές. Ε, τα email είναι επίσης πολύ σημαντικά, αλλά τις ε, τελευταίες τρεις εβδομάδες συνέβη κάτι στην Βρετανία. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ε, δεν είναι ικανοποιημένος με αυτήν την κατάσταση. Τι συνέβη λοιπόν, η Πρωθυπουργός κυρία Μέη είπε ότι η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε με ισχνή πλειοψηφία και θα πρέπει να το δεχτούμε και είπε αγαπητοί συμπολίτε, ε, δώστε μου μια ισχυρή εντολή για Brexit και θα το κάνω. Και ποια ήταν η απάντηση των Βρετανών πολιτών, ήταν ένα όχι. Βλέπω λοιπόν πόσο το θέμα είναι ανοιχτό ακόμα και στη Βρετανία. Και πρέπει να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Οποιοςδήποτε Βρετανός λοιπόν είναι εδώ πέρα καλοδεχούμενος, οπότε κύριε Βίλαμσον θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά σας στην περίπτωση που θέλετε να επανέλθετε λοιπόν και ο Τζόναθαν Κέθριτς είναι επίσης Βρετανός πολίτης και έχουμε την 1442 την αναφορά λοιπόν έχετε τον λόγο ευχαριστώ Είμαι Βρετανός που ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αναφορά μου αφορά τους πολίτες όλων των κρατών ως διεθνιστής. Εγώ θέλω να βρούμε την καλύτερη διαδικασία για την αποχώρηση οποιοδήποτε κράτους της Ένωσης. Θεωρώ πως θα πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα τα παγκόσμια και αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την ε, πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρχει δυνατότητα, να υπάρχει δυνατότητα σε μεμονωμένους πολίτε να προσβάλλουν αποφάσει που παραβιάζουν τα δικαιώματά του. Το άρθρο 50 δεν περιγράφει το πώ πλήττεται η υπηκότητα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το Brexit θα αποτελέσει δεδικασμένο για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ένα πραγματικό κίνδυνο για την αξία τη μελλοντική της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, εάν αφήσουμε να πρετανεύσει η κρατική ισχύς. Οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται μια διαδικασία εύρωστη. Η αναφορά μου ζητάει άμεση επικοινωνία και ενημέρωση όλων των πολιτών για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και μια εξήγηση των γεγονότων που θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες ε, να προσβάλλουν αποφάσεις που τους επηρεάζουν προσωπικά. Θεωρώ ότι η Ένωση θα πρέπει να διοργανώσει ακροάσεις στην Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μπορούν οι πολίτες ε, να το πώς θα Είναι ένα ηθικό και νομικό ζήτημα, αλλά αφορά και την αποτελεσματική διοίκηση, θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες και βεβαίως να υπερασπιστούμε τα όσα έχουν επιτύχει οι πολίτες. Ζητάμε λοιπόν σαφήνεια για την νομική διαδικασία, για το θέμα της ε, Ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είναι ένα ζήτημα κοινή λογική, αλλά το να καθορίσουμε το πώ θα συμβεί είναι σημαντικό γιατί έτσι θα δούμε το πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το στεγματικό δίκαιο για να επηρεάσουν οι πολίτε την διαδικασία και να μπορέσουν να προσφύγουν κατά οποιασδήποτε αδικία. Η ηθαγένεια τη Ένωση είναι επιπρόσθετη στην εθνική υπηκότητα, είναι υπερεθνική και συμπληρωματική αλλά διακριτή από την εθνική υπηκότητα. Ως πολίτης αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει σχέση μεταξύ της εθνικής και υπερεθνικής υπηκότητας, αλλά αντιλαμβάνομαι και τις διαφορές και τις εκτιμώ. Εκτιμώ τα δικαιώματα που μου δίνει η ευρωπαϊκή υπηκότητα και το ότι μπορώ έτσι να είμαι μέλος μιας ένωσης 500 εκατομμύριων ατόμων και δέχομαι την ηθική αυτή υποχρέωση συμμετοχής ε, στις ευρωεκλογέ και υπεράσπισης των επιτευγμάτων της Ένωσης. Οπότε δεν σημαίνει ότι για μένα ότι απλά εξαφανίζεται η ευρωπαϊκή ηθαγένεια όταν φεύγει ένας, ένα κράτος μέλος. Με ενοχλεί και με εκνευρίζει κάτι τέτοιο. Ειδικά όταν με απελευθερώνει από τα δέσμα του εθνικισμού. Είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Και απαιτείται νομίζω το συμβόλαιο αυτό για να τερματιστεί να υπάρξουν κάποιες διαπραγματεύσεις. Τη στιγμή που είναι όλο και ευκολότερο να, υπάρχουν, να διορθούν οι πληροφορίες και να μπορέσει ο κόσμος να πει την απόψή του, δεν είναι διαντολογικό ή λογικό ένα εθνικό δημοψήφισμα να τερματίσει την υπερεθνική ηθαγένεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ένωση, λέει πω κάθε άτομο έχει δικαίωμα να ακουστεί πριν ληφθεί ένα μέτρο το οποίο θα τον επηρεάσει προσωπικά. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να συνεργαστούμε εδώ πέρα. Οι συμμετοχικές διαδικασίες θα μπορέσουν να φωτίσουν την περιπλοκότητα και να αποκαλύψουν τις αιτίες. Ε, θα δοθεί έτσι δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες ιδέες και να υπάρξει κατανόηση μεταξύ λαών και ομάδων. Οπότε, θα ήθελα να ζητήσω η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσει ένα πρόγραμμα ακροάσεων για να ακούσει τους απλούς ανθρώπους που θα δώσουν στοιχεία για το πώς θα τους επηρεάσει η απώλεια αυτής της αγένειας. Πρέπει να είναι κάτι το επίσημο που θα έχει στόχο να συγκεντρώσει στοιχεία τα οποία θα αφορούν ε, την διαμάχη αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ιδεολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις. Ιρωνικά, ίσως το Brexit, αν γίνει όπως το περιέγραψα, θα δώσει μια ευκαιρία για μια πιο περιεκτική δημοκρατία που θα ενισχύσει την λογοδοσία και τη συμμετοχή στην Ευρώπη και θα καθορίσει θετικά την σχέση της Ένωσης με τους Βρετανούς πολίτες. Οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν το τι θα συμβεί και το δικαίωμα να προσφύγουν εάν προσβάλλονται τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας εγγυηθώ ότι εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, θα συζητήσουμε το κάθε βήμα διεξοδικά, θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Το κοινό θα μπορεί να μάθει τα πάντα. Να σας ξαναπώ επίσης ότι δεν έχουν τελειώσει τα πάντα. Υπάρχουν ακόμα δύο χρόνια, μπορούν να αλλάξουν πολλά σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν συναδέλφοι που θέλουν το λόγο. Ναι, εσείς, κύριο Σκόρμπετ, ευχαριστώ. Καμνίζω τώρα σε ευρωβουλευτής, όχι εκπροσωπώντα κάποιον αναφέροντα. Για το ότι πρέπει να ακούμε του πολίτες. Ανέκαθεν προσπαθούσαμε να το κάνουμε αυτό. Με διάφορους τρόπους. Οι περισσότερες επιτροπές μας έχουν δημόσιε ακροάσει για διάφορα ζητήματα που αφορούν το Brexit, αλλά σωστά λέει ο αναφέροντα ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και με τρόπο που θα διευκολύνει τις δυνατότητες για τους πολίτες. Και εσείς εδώ, ερχόμενος, δαπανώντας χρόνο και χρήμα, αυτό είχατε κατά νου. Αλλά να θυμόμαστε ότι πολλοί πολίτες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Πρόεδρε, δυστυχώ έχω και άλλη συνεδρίαση, οπότε πρέπει να φύγω σε λίγο. ό,τι να πω. ότι όλε αυτές οι αναφορές εξερευνούν μια οπτική γωνία συγκεκριμένη των επιπτώσεων του Brexit. Αυτές οι αναφορές είναι η κορφή του παγόβουνου και αυτό μας υποδεικνύει το εύρος και το πλάτος αυτής της υπόθεσης. Πολλοί Βρετανοί πολίτες θεωρούνται να θεωρούν ότι μπλέκονται εδώ, ότι τους αφορά αυτή η διαδικασία, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι αν παραγνωρίσουμε κάποια πράγματα αυτό θα είναι επικίνδυνο. Είναι εις βάρος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάτριτς, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση της αναφοράς σας. Θα αφήσουμε και την αναφορά σας ανοιχτή και περνάμε τώρα στον Dennis Hicks. Αναφορά 808. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ στους παρόντες. Να πω καταρχάς ότι ποτέ δεν ασχολήθηκα με την πολιτική. Είναι η πρώτη φορά επειδή έφτασα στο σημείο να απαρνηθώ το ίδιο το κοινοβουλίο μου, το εθνικό μου κοινοβουλίο μου, γιατί θεωρούσα δεν με βοηθάει πια και προσέφυγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δουλειά μου είναι το να δημιουργώ πλούτο και πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω και πολλά σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις οδηγίες κτλ. Ελπίζω βέβαια το ρίτσα ας πούμε να περιλάβει και δική μου εταιρεία, αλλά έρχομαι εδώ ως ε, μεμονωμένο άτομο για να μιλήσω στην ε, Επιτροπή σας σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε εφ' εξής. Ε, και να χρησιμοποιήσω λίγο και την ε, δημιουργία συνένεσης, λαμβάνοντας υπόψη και το δικό μου το υπόβαθρο. Θα σας μιλήσω λοιπόν σύντομα και θα ήθελα να πω τα εξή. Το πρώτο είναι ότι δεν μ' αρέσει να με χρησιμοποιούν ως διαπραγματευτικό χαρτί σε αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται. Θεωρώ ότι η ιδέα της Ευρώπης ωφελείται αν παραμείνουν οι Βρετανοί πολίτες στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα οι νέοι της Βρετανίας θα ζητήσουν την επιστροφή στην οικογένεια αυτή. Εγώ θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρήσει τον Brexit ως μια πολύ περίπτωση και μετά από αυτό να βρει έναν τρόπο ώστε να έχουμε ένα, μια γρήγορη πορεία προς μια μορφή εθνικότητας που θα περιλαμβάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο με τρόπο που θα αποφασίσουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Να σας πω δύο πράγματα για μένα. Ήρθα εδώ το 1991 στο Βέλγιο, με έστειλε η επιχείρησή μου, η εταιρεία μου. Μετά πατρεύτηκα μία Γαλλίδα της Γαλλίδας αυτής οι γονείς ήταν Πολωνοί που είχαν δραπετεύσει από την Πολωνία πριν το ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί έπρεπε να αποφασίσουν κατά πόσο θα μείναν εκεί, θα πήγαιναν στη Γαλλία, στην οικογένειά τους. Και τα παιδιά κάνουν τακτορικά και έχουν διπλή δικότητα Θα μπορούσατε να πείτε λοιπόν ότι εκπροσωπώ ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της ευρωπαϊκής ιδέας που θα μπορούσε να συναντήσει κανείς. Βλέπετε λοιπόν ποιος είμαι και καταλαβαίνετε ότι αν μπορεί να το πούνε οι διερμηνείς είμαι πώς να το πω χαμένος τελείως και τρομαγμένος μετά από όλα αυτά που συνέβησαν και ε, η πολιτική μας και ο τύπος μας επέτρεψαν τέτοιες υπεραπλουστεύσεις να καθορίσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Να προσπαθήσω να το αναπτύξω αυτό, να το εξηγήσω. Μετά το δημοψήφισμα αισθάθηκα σαν την Πολωνίδα πεθερά μου να αποφασίσω αν θα έπρεπε να δραπετεύσω ή όχι. Γιατί είχα περισσότερη περιουσία και εξάρτηση από την ε, βελγική μου σύνταξη από την Βρετανική. Ζω στην ε, Γαλλία, αλλά δυστυχώ ε, έμεινα μόνο ένα χρόνο στο, στη Βρετανία, το οποίο σημαίνει ότι έχω χάσει αυτή την συνέχεια διαμονής. Ελπίζω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω ο τελευταίος δημοκρατικός θεσμό θα αποδεχτεί ότι ο πλούστερος τρόπος για να πλήσει κανείς κάποιος αγγεμένα αυτό το δίλημα είναι το να αναζητήσει μια άλλη εθνικότητα. Αν βρείτε λοιπόν κάποιο τρόπο να πείσετε τις γειτονικές σας χώρες ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση το Brexit, τότε μπορούμε να αποφύγουμε την ε, τύχη να τον παράγοντα τύχη σε αυτή την υπόθεση. Εγώ είχα έναν παππού Ιρλανδό και διατρέχω τον κίνδυνο να έχω παιδιά με γαλλική υπηκότητα, περιουσία στο Βέλγιο και στην ε, Γαλλία με, δυνα... με ενδεχόμενο υποχρεωτική θεώρηση για να έχω πρόσβαση σε αυτά. Ήρθα εδώ και μετά το 1992 αποφάσισα να μείνω εδώ. Και το άλλο που θα ήθελα να πω, δεν ξέρω κατά πόσο νομικά είναι σωστό, παρόλο που είχαμε συζήτηση με έναν δικηγόρο σήμερα το πρωί, θεωρώ ότι να χρησιμοποιήσει αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ε, Βρετανούς ως διαπραγματικό χαρτί και αυτή, θεωρώ ότι και αυτό είναι άδικο. Νομίζω ότι έχουμε την αρχή της μη διάκρισης λόγω εθνικότητας, και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το διατηρήσει στις συνθήκες και στην ε, νομοθεσία της για πολύ καιρό μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και το λέω ως Ευρωπαίος πολίτης. Θα ήθελα να πω ότι έκανα αίτηση για εθνικότητα, για επικότητα, περίμενα τέσσερις μήνες και θα ζητήσω και μια διαπαρμονή γαλλική γιατί με ανησυχεί τόσο πολύ το τι θα συμβεί σε 1,5 χρόνο από τώρα. Αναζητώ λοιπόν οποιαδήποτε δυνατότητα για να διατηρήσω τη ζωή, τη δική μου και της οικογένειάς μου. Να πω και κάτι άλλο σε σχέση με κάποια θέματα που ακούσαμε σήμερα. Ακούμε τώρα κάποια πράγματα για αμοιβαιότητα στις διαπραγματεύσεις και αυτό με τρομοκρατεί. Και το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αρκετά καλή για να ώστε να επιτρέψει στο νέο Βασίλειο να παραμείνει στην Ένωση, τότε θα μπορούσα έτσι να καταθέσω μια σκέψη αν θέλετε οι διαπραγματεύσει αυτέ θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα ώστε οι πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου να έχουν ένα έτο στη διάθεσή του για να ενημερωθούν για τι επιπτώσει. Γιατί οι επιπτώσει τη αποχώρηση δεν είχαν συζητηθεί κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία και όπω είπαν και άλλοι συμπατριώτε μου, όταν, γίνουν γνωστέ οι επιπτώσει τη αποχώρησης τότε θα υπάρξει διαφορετική άποψη, θα αλλάξουν πολλέ απόψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κόλμπετ, έχετε το λόγο. Ναι, ε, να πω ένα τελευταίο πριν φύγω για την επόμενη συνεδρίαση. Η αναφορά αναφέρει την ε, πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία ε, σε όλα τα θέματα που αφορούν την ηθαγένεια πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο πρόβλημα. Ακόμα και αν το καταφέρουμε ακολουθώντας την αρχή του τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί, μέχρι να συμφωνηθεί, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος των διαπραγματεύσεων, πώς θα ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό οδήγησε μερικούς από εμά να ρωτήσουμε αν υπάρχει το ενδεχόμενο μιας δεύτερης συμφωνίας που θα εγκριθεί στην αρχή της διαδικασίας και να μην μας ε, κρατά σε ομοιρία η δεύτερη συμφωνία. Ο κύριος Μπαρνιέ που είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων αναφέρεται σε μία συμφωνία στον ενικό. Μία συμφωνία. Και υπάρχει λοιπόν ένα νομικό εμπόδιο. Στην ακρόαση το πρωί στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συζητήσαμε το θέμα αυτό με αρκετούς νομικούς οι οποίοι είπαν ότι εάν υπάρξει μια ικανοποιητική συμφωνία, ανάλογα με το τι θα γίνει στη συνέχεια, θα μπορούσε να υπάρξει μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και οι δύο πλευρές θα αναλάβουν, θα υποσχεθούν να εφαρμόσουν αυτά που θα συμφανηθούν, ανεξάρτητα με το πώς θα, θα πάνε οι διαπραγματεύσεις. Και αυτό πιστεύω πως αξίζει να το επιδιώξουμε και εδώ και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί θα μας βοηθούσε, θα βοηθούσε τους πολίτες να αποκτήσουν μια κάποια ασφάλεια μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη, αλλά πραγματικά πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ. Σας εγγυώμαι κύριε Χίξ ότι αυτά που αναφέρατε είναι ουσιαστικά, είναι πάρα πολύ σημαντικά, βασικά. Και για μας είναι πολύ σημαντικό, είναι η ουσία του τι κάνουμε. Δεν ε, προσπαθούμε εδώ να αλλάξουμε ή να διορθώσουμε μία απόφαση που θεωρούμε λάθος. Δεν προσπαθούμε να αντιστρέψουμε το αποτέλεσμα. Όπως είπα, αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο οι Βρετανοί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χίξ. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Μετά, Έχουμε την επόμενη αναφορά. «832». Ο αναφέρον δεν είναι εδώ για να την παρουσιάσει ο ίδιος. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην Λαουραντή Λεντίτε και την Εύα Μαρία Πορκέβα για τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Θα μας ε, παρουσιάσετε κάποιες από αυτές τις... Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την ε, πρόσκληση και την δυνατότητα να παρουσιάσουμε την δουλειά μας. Είναι τιμή και πολύ περισσότερο το ότι την παρουσιάζουμε ε, παρουσία πολιτών που επηρεάζονται άμεσα από το Brexit και πολίτες ε, ε, τα δικαιώματα των οποίων έρευνουμε εδώ και καιρό. Εγώ και οι συναδελφός μου δουλεύουμε στην υπηρεσία ερευνών του Κοινοβουλίου και παρέχουμε ερευνά σε επιτροπές και βουλευτές πέρα από τις εμπιστευτικές έρευνες κάνουμε και δημόσιες μελέτες όπως αυτή εδώ. Αυτή δεν έχει δημοσιευτεί, θα δημοσιευτεί όμως τις επόμενες ημέρες και καλύπτει τις προτεραιότητες της πρώτης φάσης ε, του Brexit, όπως είπε ο κ. Κόρμπετ, υπάρχουν δύο φάσεις. Εμείς καλύπτουμε τις προτεραιότητες για την πρώτη φάση, όχι μόνο τα δικαιώματα της ηθαγενείας αλλά και τα ζητήματα εγκατάστασης, τα οικονομικά και το πιθανό σκληρό σύνορο μεταξύ Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας. Τώρα θα μείνουμε στα της υπηκότητας. Λοιπόν, εστιάζουμε πάρα πολύ βεβαίως στην θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις προτεραιότητες και ασχολούμαστε και με τις συνέπειες της μη συμφωνίας Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ερμηνεία ή να λάβουμε υπόψη κάποια άλλα σενάρια πιθανών συμφωνιών. Οπότε θα δώσω τώρα τον λόγο στην συνάδελφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε τα αποτελέσματα των έρευνών μας για τα δικαιώματα των πολιτών στις διαπραγματεύσεις για τον Brexit όπως υπόθηκε ήδη. Όπως γνωρίζουμε το Συμβούλιο ανέκανε τις κατευθύνες γραμμές στα τέλη Απριλίου που παρουσιάζουν μια λεγόμενη σταδιακή προσέγγιση Δηλαδή θα έχουμε μια πρώτη φάση που θα έχει στόχο την απεμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου και το να υπάρχει κάποια βεβαιότητα για τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επίσης κάποιες κατευθυντήρες γραμμές που αναφέρουν κάποιες προτεραιότητες για αυτή τη φάση, την πρώτη φάση, που περιλαμβάνουν και τις ε, προτεραιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αυτές είχαν αναφερθεί στο ψήφισμα της 5ης Απριλίου και περιλαμβάνουν, όπως είπε η συνάδελφος, τα δικαιώματα των πολιτών, οικονομικές υποχρεώσεις, συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Ε, τα, από τα ζητήματα αυτά σήμερα καλύπτουμε μόνο τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και τα δικαιώματα της ελευθερής μετακίνησης. Η μεταχείριση και κοινωνική ασφάλιση δηλαδή εγώ θα καλύψω τα δικαιώματα παραμονής και η συνάδελφος μετά θα πει δύο λόγια για την ίση μεταχείριση και την κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή θα πούμε λίγα λόγια για το πώς έχει το τρέχον νομικό πλαίσιο, ποιες είναι και θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες και ε, είναι δύσκολο να ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά βεβαίως μπορούμε να δούμε πιο προσεκτικά την θέση της Ένωσης που έχει παρουσιαστεί τώρα σαφώς στις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου και στο έγγραφο εργασίας της Κομισιόν. Μάλιστα. Λοιπόν, ήδη υπόθηκε και γνωρίζω ότι... Εντάξει, είναι γνωστό υπάρχει ο παράγωγος χαρακτήρας της ε, κοινοτικής υπηκότητας, δηλαδή πρέπει κάποιος να είναι υπηκός κράτους μέλους για να έχει κοινωνική, κοινοτική ηθαγένεια. Και έχουμε άρα τα διάφορα επιχειρήματα που ακούστηκαν, τα οποία είναι υπέρ μιας ε, κάποιας μορφής ε, της ε, κοινοτικής ηθαγένειας διαφορετικής ε, με μεγαλύτερη συμπερίληψη. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το ε, χειρότερο πιθανό σενάριο, δηλαδή τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία και δεν υπάρξουν άλλες μονομερείς εγγυήσεις και παραχωρήσεις. Τι σημαίνει αυτό. Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είναι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους θα είναι πλέον υπήκοοι τρίτης χώρας όσον αφορά το κοινοτικό κεκτημένο και θα ισχύει το κοινοτικό δίκαιο συν το εθνικό δίκαιο περί μετανάστευσης ε, της ε, χώρας όπου κατοικούν. Τι σημαίνει αυτό όταν λέμε κοινοτικό κεκτημένο για υπηκόους τρίτων χωρών. Παραδείγματος χάρη ε, η οδηγία περί μακροχρόνιας παραμονής, η οδηγία της μπλε κάρτας για ερευνητέ και φοιτητέ υπηκόους τρίτων χωρών και τα λοιπά. Για τους πολίτες των 27 η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική με την έννοια ότι δεν θα χάσουν το καθεστώς του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά σαφώς ε, ε, εφόσον κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υφίστανται μετά τις ε, εθνικές διατάξεις περί μετανάστευσης ε, και αυτό σημαίνει και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί και Βρετανοί και Ευρωπαίοι πολίτες προσπαθούν ε, να αποκτήσουν την υπηκότητα της χώρας διαμονής. Είδαμε πριν από λίγες μέρες η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των Βρετανών που ηρανυπηκότητα τριπλασιάστηκε, υπερτριπλασιάστηκε το 2016. Και νομίζω αυτό αφορά και κάτι το οποίο είπε ένας εκ των αναφέροντων. Δηλαδή αυτό κάνουν τώρα πολλοί πολίτες δεδομένης της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν. Η μελλοντική λοιπόν συμφωνία έχει μεγάλο ρόλο για τα δικαιώματά τους. Μεγάλη σημασία όπως είπαμε, αν δεν υπάρχουν μονομερείς εγγύσει και τα κράτη-μέλη ε, μπορούν μεταξύ άλλων να πούν ότι θα είμαστε πιο επίοικείς ε, στους όρους ε, που θα επιβάλλουμε π.χ. για την πολιτογράφηση. Οπότε, ποια είναι η θέση της Ένωσης τώρα που έχει μπει επιτάπητος με ξεκάθαρους όρους. το έγγραφο εργασία της Κομισιόν. Τι θέλουν τα έγγραφα αυτά. Πρώτα απ' όλα έχουμε το καθεστώς και τα δικαιώματα τα οποία θα προκύπτουν από την πράξη απόσυρσης ε, σύμφωνα με την οδηγία αυτό θα περιλαμβάνει και δικαιώματα που θα προκύψουν αργότερα π.χ. συντάξεις δικαιώματα τα οποία είναι τώρα στην διαδικασία θεμελίωσης π.χ. δικαίωμα παραμονής που θα πρέπει να μπορεί να αποκτηθεί και μετά την ημερομηνία αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπό τους σημερινούς όρους και θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τους πολίτες των 27 στη Βρετανία την ημερομηνία ε, αποχώρησης ε, και τους Βρετανούς ε, στις 27 χώρε. τα 4-5 εκατομμύρια ανθρώπους δηλαδή και θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής για τα δικαιώματα αυτά ε, για όλη την ε, ζωή των ενδιαφερομένων. Και η Κομισιόν λέει ουσιαστικά ότι ε, θέλουμε να έχουμε λίγο πολύ το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως θερμινεύει το δικαστήριο. Οπότε ερχόμαστε στο επόμενο ερώτημα. Ποιο είναι το τωρινό επίπεδο προστασίας. φαίνεται ότι πέρασα πάλι κάποια διαφάνεια. Εντάξει, δεν θα αναφέρω λεπτομέρειε όλε τι κατηγορίες της διαφάνεια Ήμουν εδώ και το πρωί και ξέρω ότι καλύφθηκαν ήδη πολλά από αυτά τα σημεία. Παρ' όλα αυτά, με πω τα Τι γίνεται την προστασία το δικαιωμάτων των πολιτών. Είχαμε την οδηγία που καλύπτει τα δικαιώματα των πολιτών και τις προϋποθέσεις διαμονής που εξαρτώνται από τους εμπλεκόμενους αυτοπασχολούμενους, οικονομικά μη ενεργούς, εργαζόμενους κλπ. Το να εργάζεται κανείς επαρκεί συνήθως και το δικαστήριο ήδη στην πρώιμη νομολογία του ξεκάθαρα είπε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την έννοια πανευρωπαϊκά γιατί δεν επαρκεί να έχουμε γενναιόδορες ορισμούς ή διατάξεις αν μετά μπορούν να ερμηνευτούν αυτές περιοριστικά από τις χώρες μέλη. Εργαζόμενος λοιπόν είναι το, το κάθε άτομο που έχει μία δραστηριότητα απασχόλησης. και κατά πόσο εργάζεται λίγες ώρες ή η αμοιβή του είναι χαμηλή, αυτό δεν έχει τόση σημασία. Αυτό τι σημαίνει. Ακούσαμε το πρωί ότι κάποιες χώρες εφαρμόζουν κάποια κατόφλια ελάχιστου εισοδήματο ή ορών εργασίας ανά εβδομάδα. Δεν το βλέπει έτσι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πάλι μια συμφωνία αποχώρησης θα μπορούσε να είναι πολύ γενναιόδορη προς τους εργαζόμενους αν οριστεί περιοριστικά και να ευνοήσει λίγους. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τώρα θα πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε για διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι ο ορισμό του εργαζόμενου. Η Κομισιόν λέει είναι ότι ότι είναι αυτός ο ορισμός του δικαστηρίου. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις άτυπες μορφές απασχόλησης, γιατί έχουμε σε αυτά τα άτομα να διατρέξουν κινδύνους. Για τις άλλες κατηγορίες, και ιατρική περίθαλψη και ασφάλεια ασθένειας. η πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι αποδεκτή από τις Βρετανικές Αρχές. Η Κομισιόν το 12 ξεκίνησε μια διαδικασία παράβασης για αυτό το ζήτημα που επιβεβαίωσε ως υποεξέλιξη η Κομισιόν το 16 αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώ ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης γνωρίζοντας δηλαδή ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αποχώρησης, γιατί θα μπορούσε να έχει πολύ αρνητικέ επιπτώσεις σε αυτούς που χρησιμοποίησαν ακριβώς τις ε, συνθήκες ελεύθερης κυκλοφορίας. Για τα μέλη των οικογενειών. Τα μέλη των οικογενειών ανεξαρτήτως υπηκότητας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματα που προβλέπουν οι συνθήκες. Θα πρέπει να δούμε όμως και το εξής. Υπόκειται σε πιο αυστηρές προϋποθέσεις οι πολίτες των χώρων της Ένωσης όσον αφορά τα θέματα επανένωσης. Ανεξάρτητα από αυτά που προβλέπουν οι συνθήκε όσο γενναιόδορε και να είναι. Και μάλιστα χθε το κοίταζα, αυτή η οδηγία σε σχέση με την εφαρμογή της ε, υπηκόου τρίτων χωρών και για το τι θα μπορούσαν να χάσουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες Πράγματι, στα πλαίσια της επανένωσης επιτρέπει στις χώρες μέλη να ζητήσουν την ύπαρξη σταθερών και τακτικών πόρων. Ας πούμε, επιτρέπεται στις χώρες μέλη να επαληθεύσουν κατά πόσο υπάρχει κατοικία αρμόζουσα και συνθήκες ένταξης όσον αφορά τη γλώσσα κλπ. Οπότε, σε περίπτωση μη συμφωνίας, οι πολίτες της Ένωσης θα χάσουν πολλά, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικογενική επανένωση και τα μέλη των οικογενειών τους. Δεν θα μιλήσω για την επόμενη διαφάνεια, για τα τυπικά και τα γραφειοκρατικά ζητήματα και θα δώσω τώρα το λόγο στην συνάδελφο που θα μιλήσει για θέματα ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης. Είπαμε, ναι, ότι το δικαίωμα διαμονής δεν είναι σημαντικό επειδή επιτρέπει να πας να ζήσεις σε μια άλλη χώρα, είναι σημαντικό λόγω των παρελκομένων του. Και ένα από τα δικαιώματα αυτά είναι το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Ένωσης, το οποίο σημαίνει ότι ένας πολίτης της Ένωσης πάει σε μια άλλη χώρα μέλος και αποφασίσει να σπουδάσει, να δουλέψει, να μείνει ο συνταξιούχος, σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διακρίσεων. Και δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να είναι αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης λόγω υπηκότητας, όπως ας πούμε όταν πάτε ας πούμε, να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες και σας λέω θα πρέπει να πληρώσετε περισσότερα επειδή δεν είστε Βρετανός υπήκος και βλέπουμε ότι ήδη συμβαίνει από ό,τι φαίνεται στον βρετανικό τύπο. Η επίπτωση λοιπόν αυτής της διάταξης είναι πολύ πιο αρνητική για τις πολίτες της Ένωσης από ότι για τους Ας πούμε μια περίπτωση ενός ε, φοιτητή που θέλει να σπουδάσει σε διαφορετική χώρα μέλος και όχι στην δική του και μπορεί να υπάρξει αυτή η απέτηση ας πούμε για απολυτήριο λυκείου από την ίδια χώρα το οποίο βεβαίως αποκλεί τους μη υπηκόους. Γι' αυτό και το οποίο είναι μια διάκριση. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν στο έγγραφό τη λέει ότι αυτό πάνω στο οποίο θα επικεντρωθεί η Κομισιόν είναι η διασφάλιση της ε, ίσης μεταχείρισης. Ίση μεταχείριση μεταξύ πολιτών Βρετανίας και πολιτών 27 χωρών της Ένωσης. Βέβαια, έχουμε και άλλες κατηγορίες πολιτών στην Ένωση πολίτες οι οποίοι έχουν δικαιώματα υπό την Βρετανική νομοθεσία, αλλά δεν θα επικεντρωθεί βεβαίω ότι πραγματευτεί και η κοινότητα σε αυτό, αλλά ίση μεταχείριση για τους πολίτες ενός και όχι για τους πολίτες τρίτων χωρών. Ίση μεταχείριση βεβαίω και των Βρετανών στην Ένωση και μεταξύ βεβαίως των πολιτών των 27 χωρών της Ένωσης ως εφαρμογή αυτής της αρχής της ενότητας που εξέφρασαν οι τελευταίες γραμμές του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ότι δηλαδή δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις χωριστές μεταξύ μεμονωμένων χωρμερών και Βρετανίας αλλά θα γίνουν υπό τον διαπραγματευτή δηλαδή την Κομισιόν στο όνομα των χωρών μελών. Βεβαίως, ξέρουμε ότι στη Βρετανία για κάποια δικαιώματα που ήδη προϋπήρχαν για το δικαίωμα ταξιδιού ή μετακίνησης, δηλαδή στην περίπτωση της Ιρλανδίας, ε, το σύνορο με τη Βρετανία, οι Ιρλανδοί πολίτες έχουν όμως και άλλα δικαιώματα. Θέλουμε λοιπόν την ίση μεταχείριση για όλους τους 27. Οπότε αυτό θα πρέπει να αφορά και τους πολίτες της Ιρλανδίας. Το οποίο σημαίνει ότι η νομοθεσία θα πρέπει να μείνει ως έχει. Και κάτι άλλο σε σχέση με την ίση μεταχείριση. Αυτό θα πρέπει να αριθμιστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την ερμηνεία του, δικαστηρίου μετά τη συμφωνία. Το πάγωμα της ίσης μεταχείρισης σημαίνει αφενός ότι αν μελλοντικά έχουμε μια δευτερεύουσα νομοθεσία με περιορισμούς στην ίση μεταχείριση, αυτό καταρχάς δεν θα αφορά τους πολίτες της Βρετανίας που ζουν στην Ένωση ή αντίστροφα αν αυτό βέβαια δεν ε, είναι αντικείμενο συμφωνία στα πλαίσια διαπραγμάτευση. Επίση, για την κοινωνική πρόνοια και ο αντίστοιχο ε, συντονισμό δεν το ονομάζουμε κοινωνικά δικαιώματα, αλλά μιλάμε για κοινωνική πρόνοια. Γιατί είναι κάπω έτσι υψοκίνητο ο όρο κοινωνικά δικαιώματα. Γιατί είναι σημαντικό. Επειδή πραγματικά αντανακλά την εφαρμογή τη αρχή τη ίση μεταχείριση. Δηλαδή, αν πάτε να δουλέψετε σε άλλη χώρα μέλο, Βεβαίω έχετε το δικαίωμα εργασία εκεί. Αν όμω δεν έχετε τα ίδια δικαιώματα με του υπηκόου εκείνη τη χώρα πιθανώ να μην πηγαίνατε. Αυτό τι σημαίνει τώρα. συντονισμό θεμάτων κοινωνική πρόνοια, καταρχά, όπω λέγαμε, είσαι μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων από την Ένωση και επικών της χώρας. Επίσης, το ότι εφαρμόζεται μόνο και ισχύει μία, μία νομοθεσία. Δηλαδή αυτοί που έχουν πληρώσει τις ε, εισφορές τους σε μία χώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει, από το οποίο συνοδεύεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δηλαδή ισχύει και εφαρμόζεται η μία νομοθεσία. Μετά, προσθήκη περίοδων διαμονής και κοινωνικά επιδόματα. Αυτό που ζητούν είναι να έχει εισφέρει κανεί στα δημόσια ταμεία συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η δυνατότητα προσθήκη σημαίνει ότι αν έχετε εργαστεί σε κάποια άλλη χώρα, α πούμε, έξι μήνε, μετά πάτε σε άλλη χώρα μέλο και δουλεύετε άλλου έξι μήνε, φανταστείτε ότι αυτή η χώρα λέει ότι για να σου δώσω πούμε, επίδομα ανεργία, πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον για ένα έτος. Αυτή λοιπόν η αρχή τη προσθήκη ή τη ισόρευση, επειδή ακριβώ αφορά διαφορετικέ χώρε μέλη, αυτέ οι χρονικέ περίοδοι προστίθενται, οπότε εσύ έχει δικαίωμα για επίδομα ανεργία. Οπότε είναι πολύ πρακτική η τη ισορρευση επειδη ακριβω αφορα διαφορετικε χωρε μελη αυτε οι χρονικε περιοδοι προστιθενται οποτε ακριβώ των γενικών δικαιωμάτων. Εξαγημότητα αν έχετε εσείς μια σύνταξη, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται να μείνετε στη χώρα σας, κάτι το οποίο κάνουν πολλοί πολίτε της Βρετανίας και αποφάσισαν πραγματικά να πάνε πούμε, στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Και μπόρεσαν να λάβουν τις ε, συντάξει τους εκεί, σε αυτές τις χώρες. Οπότε, να δω την επόμενη διαφάνεια δικαιώματα των εργαζομένων. Όπως λέγαμε προηγουμένως, ή μεταχείριση σε σχέση με θέματα αμοιβών, σχετικών εργασία κλπ. Επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας στην χώρα μέλος όπου εργάζονται, επιδόματα ασθένεια, επιδόματα ανεργία, οικογενειακά επιδόματα, όλα αυτά θα πρέπει να είναι ισότιμα με αυτά που λαμβάνουν οι υπηκοί αυτές της χώρας. Τώρα μετά το Brexit ε, πρέπει να πούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχαν κάποια εσωτερικά επιδόματα στις επιχειρήσεις. Ας πούμε ε, πιστώσεις που διδόταν στους εργαζομένους ή κάποιες άλλες παροχές που αντιστάθμιζαν τα χαμηλά εισοδήματα, τις χαμηλές αμοιβέ. Οι χαμηλέ λοιπόν αμοιβέ ε, συμπληρώνονταν από αυτά τα επιδόματα. Τώρα τι γίνεται. Δεν αφορούν οι εισφορέ σε δημόσια ταμεία, αλλά δίδονται ανάλογα με το εισόδημα του καθενός για τη διαβίωσή τους. Υπό την Βρετανική λοιπόν νομοθεσία αυτά τα επιδόματα δεν δίδονται σε υπηκόους τρίτων ε, χωρών. Στους πρώτες ένωσης ναι, αλλά αν γίνουν πολίτες τρίτων χωρών, οι πολίτες ενώσεις υπό την Βρετανική νομοθεσία, τότε δεν θα έχουν δικαίωμα αυτών των επιδομάτων και θα δεχτούν διάκριση σε σχέση με τους υπηκούς της Βρετανίας. Μετά, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά αυτών των πολιτών. Η ίδια με αυτή που αφορά τα παιδιά των υπηκών εκεί της χώρας. Μετά, παιδικά επιδόματα, κάτι το οποίο συζητήθηκε. Θυμάστε, ο Κάμπερο το είχε διαπραγματευτεί αυτό με την Ένωση, ώστε να μπορέσει τέλο πάντων, είχε πει αυτός, να κάνει εξαρτία υπέρ της παραμονής δέχτηκε πολλές επικρίσεις το γεγονό ότι αυτές, αυτά τα, παιδικά επιδόματα μπορούν να εξαχθούν αν εργάζεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, έστω δηλαδή και αν τα παιδιά σα παραμένουν στη χώρα προέλευση, ζουν στη χώρα προέλευση και σε αυτή την περίπτωση δικαιούστε παιδικά επιδόματα. Επειδή απολαμβάνουν το ίδιο κοιμάτων που απολαμβάνουν οι Βρετανοί εργαζόμενοι. Και αυτό ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και είναι κάτι για το οποίο αναμένουμε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία υπό την Βρετανική Νομοθεσία και αυτό θα τροποποιηθεί, θα αλλάξει. Άνεργοι. Επιδόματα, συμπλήρωση χρονικών περιόδων και επιδόματα τα οποία αφορούν περιόδους άνω των έξι μηνών, ώστε να ζητήσουν ε, εργα, εργασία σε άλλη χώρα μέλος. Σε περίπτωση δεν υπάρξει συμφωνία και αυτό θα εξαλειφθεί. Καταλήγοντας κάποιες άλλες κατηγορίες, συνταξιούχοι, τα χρόνια εργασίας, και συμπλήρωσή τους. Αν έχετε εργαστεί, ας πούμε, ως πολίτες Ένωσης σε τρεις διαφορετικές χώρες μέλη, για ένα χρόνο τουλάχιστον, ε, δικαιούστε τρεις συντάξεις. Αν όμως έχετε εργαστεί, ας πούμε, έξι μήνες σε μια χώρα μέλος, δεν έχετε δικαίωμα σε συνταξή του σε αυτή τη χώρα. Θα προσθεθούν όμως αυτές οι χρονικές περίοδοι ώστε να μην χάσετε ακριβώ τι εισφορέ σα και να, να συνεισφέρουν στο ύψο τη σύνταξη. Κάτι άλλο που αφορά του κανόνε συντονισμού είναι η περίθαλψη. Η περίθαλψη ίδια δεν εξάγεται, παρέχεται στη χώρα διαμονή, όμως η χώρα διαμονή αποζημιώνεται για την περίθαλψη η οποία παρέχεται από την χώρα η οποία καταβάλει τη σύνταξη. Αυτά που ακούσαμε λοιπόν για τους ε, Βρετανούς ταξιούχους στην Ισπανία που περιθάπτονται και αποζημιώνεται μετά η Ισπανία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, υπάρχει επίκριση για το σύστημα αυτό. Υπάρχουν κριτικές επειδή η Ισπανία δεν αποζημιώνει το πραγματικό κόστος, αλλά χαμηλότερο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, το πώς οι χωρε μέλη προετοιμάζονται ακριβώς για τις επιπτώσει του Brexit, η τονή κυβέρνηση της Ισπανίας ήδη ανακοίνωσε ότι ίσως να υπάρξει, ότι θα υπάρξει αλλαγή στην εμφανισία, Δηλαδή, στη, στο μέλλον, οι συνταξιούχοι θα έπρεπε να έχουν ιδιωτική ασφάλεια για να τύχουν περίθαλψη στην Ισπανία. Για την περίθαλψη πρέπει να πούμε επίσης ότι έχουμε σε επίπεδο ένωσης την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας που παρέχει δυνατότητα στους πολίτες της Ένωσης όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη. Και αυτό θα χαθεί αν δεν έχουμε συμφωνία. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μας και βλέπουμε σε γενικές γραμμές ότι οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές για τους υπηκόους της Ένωσης. Και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς η προσπάθεια για τη διατήρηση των δικαιωμάτων όσο έχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση της μελέτης. Είναι πραγματικά πολύ καλή επαγγελματική δουλειά και πιστεύω πως θα μας φανεί πολύ χρήσιμη. Θα παρακολουθούμε λοιπόν και εμείς ε, τις εξελίξεις και σημειώνουμε να ξέρετε τα όσα ακούσαμε. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Με ενημέρωσαν ότι η αναφορά 879 της κυρίας Σοφιλέιτον δεν μπορεί να παρουσιαστεί. Λάβαμε μια επιστολή από τον κύριο Λέιτον. Και γι' αυτό που μας εξηγεί σχετικά και θα περάσουμε στην επόμενη αναφορά 0393 του 2019 του TJ δεν ξέρω καν αν πρόκειται για γυναίκα ή για άντρα που υπέβαλε την αναφορά, αλλά θα έπρεπε να είναι εδώ. Ο κύριος TJ λοιπόν και θα του δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αναφορά αυτή αφορά τις συντάξεις για άτομα όπως εμένα που εργάστηκαν και στη Γαλλία αλλά και στην Βρετανία. Αναφέρεται το κείμενο ότι καταβάλλεται η Βρετανική Σύνταξη πανεθνικά. Παρ' όλα αυτά η αύξηση στη σύνταξη θα δοθεί μόνο αν διαμένεται αν διαμένετε μόνο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στο Γιβραλτάρ ή την Ελβετία. Ή μια κάποια άλλη χώρα που έχει κάποια συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης με το Ηνωμένο Βασίλειο που μπορεί να, εσύ, να συμπολιστεί στη σύνταξη και να καταστεί επιλέξιμος ο πολίτης. Και ο, ο γυρίζει στα γαλλικά. Λοιπόν, υπάρχει η βασική κρατική σύνταξη, η οποία αυξάνεται κάθε χρόνο ανάλογα με το τι είναι πιο υψηλό. Τα ε, έσοδα, οι τιμές, το η ποσοστία αύξηση στις τιμές ε, όπως τη μετρά ο δείκτης ε, τιμών των καταναλωτικών προϊόντων τουλάχιστον 3%. Έτσι αναφέρει το κείμενο, έτσι έχει κατάσταση στην Μεγάλη Βρετανία προς το παρόν. Θέλω τώρα σύντομα να σας παρουσιάσω τα κύρια σημεία της αναφοράς. Παντρεύτηκα το 1973 μια Γαλλίδα υπήκο το 1973, τη ίδια χρονιά δηλαδή που προσχώρησε στην Ένωση τότε κοινότητα η Βρετανία. Από το 1978 και μετά ε, η λέξη δηλαδή ήταν Ευρώπη. Εγώ είχα εργαστεί λοιπόν και στην Βρετανία και στην Γαλλία και όλες οι συμβάσεις εργασίας μου αφορούσαν μια αμοιβαιότητα μεταξύ παρόχου και πελατών. Αλλά αυτό δεν ισχύει για την συνταξιδότησή μου. Και υπάρχει ένας υπαρκτός κίνδυνος, γιατί πραγματικά μετά το Brexit θα αλλάξουν οι υπολογισμοί μόνο των, του ύψους συντάξεων και δεν θα σε εμποδίσει τίποτα. Σύμφωνα με την ε, Guardian, είμαστε 1.200.000 υπήκοοι Βρετανοί που ζουν στην Ευρώπη και η λέξη δεν είναι υπήκοοι. Πολίτες. Η Ευρώπη λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει και αυτό ακριβώ κατέθεσε αυτή την αναφορά. Ελπίζω να τύχω της υποστήριξή σας και ότι θα την ε, λάβετε υπόψη σας στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Επειδή ακριβώς οι αναφορές χρειάζονται και στη συνέχεια τους ε, υπογραφές, αν με βοηθήσετε θα προσπαθήσω να το πράξω. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ένωσης. Δεν θα πρέπει που δεν να να παγώνει ή να μειώνεται η Βρετανική σύνταξη βάσει αυτών των διακρίσεων. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν θα πρέπει να, να τιμήσει τις δεσμεύσεις του όσον αφορά τους Βρετανούς που διαμένουν εκτός Ενωμένου Βασιλείου αλλά στο εσωτερικό της Ένωσης και σε περίπτωση μη ε, εφαρμογής μετά το Brexit θα πρέπει να λάβει τις δεσμεύσεις της Βρετανίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν θα συνταξιωθούν αυτοί οι πολίτες, οι Βρετανοί. Οι πολίτες λοιπόν, οι εργαζόμενοι, αυτοί που αναφέρατε προηγουμένως, οι πολίτες λοιπόν έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στις ταξιδοτικές τους εισφορές. Τώρα η Βρετανική κυβέρνηση με τη σειρά τη έχει την υποχρέωση να καταβάλει συντάξεις. Πρέπει λοιπόν αυτή η υποχρέωση να μην αλλάξει κατά διάρκεια της περίοδου συνταξιοδοτήσεως. ανεξάρτητα από ποια κυβέρνηση θα υπάρχει στην Βρετανία. Ήδη εξάλλου σήμερα το απόγευμα μιλήσαμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Βρετανία αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ένωση και 500.000 συνταξιούχοι όμως έχουν την υποχρέωση να προστατεύσουν τις συντάξεις τους. Γιατί ξα... πρέπει να σας ότι το μόνο έσοδο για τους συνταξιούχους είναι η σύνταξη. Να σας δώσω και δύο παραδείγματα. Έχουμε αυτούς που είτε μέσα στην Ευρώπη για πάνω από 15 χρόνια Αυτοί δεν μπορούσαν να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Ήδη είχαμε μια απώλεια της τάξεως του 11% μετά από την μείωση της οτιμίας της λίρας σε σχέση με το ευρώ. Αλλά εντάξει, επιλέξαμε να ζήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δικό μας πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που λαμβάνετε, που θα λάβετε υπόψη την αναφορά μου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον Brexit και θα ακούσαμε προσοχή της απόψης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η αναφορά έγινε παραδεκτή και θα ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το περιεχόμενο. Γι' αυτό ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Ε, κύριε Κέρτον Ντάρλινγκ, ευχαριστώ. Ως ε, συνέχεια της αναφοράς του κύριου Χίξ, θα ήθελα να πω ότι εδώ φαίνεται από προσωπικές μελέτες με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς ε, συμβαίνει και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις ζωές ε, των ε, ανθρώπων εάν δεν επιτευχθεί μια καλή συμφωνία, όχι μια οποιαδήποτε συμφωνία. Μια συμφωνία που δεν θα μειώσει τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν θα τους απογοητεύσει δεν θα αλλάξει τη ζωή τους. Ε, μια ζωή την οποία έχτισαν βασισμένη στις ελευθερίες που απολαμβάνει ένας Ευρωπαίος πολίτης. Και θα ήθελα λοιπόν να πω στου αναφέροντες ότι να είστε σίγουροι όταν θα ε, περάσουμε στις ε, συζητήσει για την θέση του Κοινοβουλίου θα χρησιμοποιήσουμε τις δικέ σα περιπτώσει, τι δικέ σα αναφορέ, έτσι ώστε να δώσουμε συγκεκριμένα αυτά παραδείγματα. Διότι όταν αναφερόμαστε σε νούμερα είναι απρόσωπο, ξέρετε. Το 4,5 εκατομμύρια ε, δεν μας λέει κάτι, αλλά αυτά τα 4,5 εκατομμύρια είναι 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, 4,5 εκατομμύρια ιστορίες. Σημαντικό λοιπόν είναι αυτές οι δικές σας ιστορίες να ε, λάβουν σάρκα και ωστά και να τις χρησιμοποιήσουμε όταν θα ε, συγγράφουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, τη θέση του Κοινοβουλίου. Αναφέρθηκα ήδη ότι έγινε και μια συζήτηση στην Επιτροπή των Σταγματικών Υποθέσεων για τα Δικαιώματα των Πολιτών και στην ακρόαση που έγινε ε, την κοινή ακρόαση των Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της δικής μας, ο Κίφερ Χόφστατ είπε πως ε, μιλώντας εκ μέρους του Κοινοβουλίου δεν θα δεχόταν μία συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, Μεγάλη Βρετανία και το Ηνωμένο Βασιλείο, η οποία δεν θα δεν θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι και η δική μας ε, θέση, η δική μας στάση δείχνει το πόσο δεσμευόμαστε για να απολαμβάνετε τα δικαιώματά σας και στο μέλλον. Είναι δικαιώματα τα οποία πιστεύω πως όλοι θα έπρεπε να έχουμε και εγώ και εσείς πρέπει να μας εγγυηθούν τουλάχιστον αυτό. Και ο επικεφαλής της αντιπραγμάτευσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε σαφέστατα κατά τις επαφές του με ε, τους ε, υπόλοιπους διαπραγματευτές ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι να προστατεύσει τους πολίτες και τα δικαιώματά τους. Τώρα λοιπόν πρέπει να μπούμε στις λεπτομέρειες, να δούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Γι' αυτό οι δικές σας αναφορές θα μας χρησιμεύσουν έτσι ώστε να μπορέσουμε βασισμένοι σε αυτές να κάνουμε τις ε, κέρυες ερωτήσεις στην άλλη πλευρά. Και σήμερα, σήμερα το απόγευμα είχαμε την πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου με την ε, ομάδα παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς είμαι εδώ και δεν μπορούσα να πάω. Αλλά αυτή η ομάδα αποτελείται από ευρωβουλευτές και εξετάζει τι ακριβώς ε, συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις. Οι αναφορές σας λοιπόν θα μας δώσουν, αν θέλετε, τη δυνατότητα να μπούμε σε λεπτομέρειες, να ρωτήσουμε συγκεκριμένα πράγματα κατά τις διαπραγματεύσεις. Πώς ε, σκοπεύετε να λύσετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Γιατί θα κάνετε αυτό που θα κάνετε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό εσείς να υποβάλλετε αναφορές, να θίγετε αυτά τα θέματα, διότι πραγματικά βοηθά τους ευρωβουλευτές στη δουλειά τους, μας βοηθά να ε, ερευνούμε, να εξετάζουμε και... Ε, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά σας και να φροντίσουμε να μην τα χάσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παραμένει νυχτή και αυτή η αναφορά και θα ενημερώσουμε την Κομισιόν για το περιεχόμενο. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα αφορά το πρόγραμμα Erasmus Plus. Ε, πάλι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Brexit και 10.000 άτομα υπέγραψαν την αναφορά. Πρόκειται για την 174 του 2017, έχετε τον λόγο. Γεια σας. Έχω έρθει σήμερα εξ ονόματος των νέων φιλελευθερών για να παρουσιάσω την ε, αναφορά μας. Εμείς ζητάμε, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Erasmus Plus. Εδώ και 30 χρόνια το πρόγραμμα Erasmus Plus έχει εμπλουτίσει τις ζωές των φοιτητών και των νεαρών μέσω των ανταλλαγών. Δημιουργεί τις πανεπιστημιακές και πολιτιστικές εκείνες ανταλλαγές που εμπλουτίζουν τη μάθηση η οικονομική στήριξη του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα σε νέους να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η απόδοση του Ηνωμένου Βασιλείου αυξάνεται συνεχώς. Είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους προορισμούς του Erasmus Plus και πάνω από 200.000 Βρετανοί φοιτητές ε, και σπουδαστές έχουν πάει στην Ευρώπη. Εμείς ε, θεωρούμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να παραμεριστεί το Erasmus Plus στις διαπραγματεύσεις και οι νέοι σε ολόκληρη την Ευρώπη θα τιμωρηθούν για τις αποφάσεις των μεγαλύτερων γενναίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 75% των νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισαν να παραμείνουν στην Ένωση. Όπως ακούσατε σήμερα, πολλοί από εμάς έχουν πολυεπίπεδες ταυτότητες. Θεωρούμε αυτούς Βρετανούς και Ευρωπαίους και Άρα το να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απειλή και κατά της ταυτότητάς μας ως παιδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εγώ άρχισα να σέβομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ νωρίς ε, στο σχολείο. Παίζαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίναμε να διαπραγματευόμαστε και να συζητάμε με μαθητές από όλο και την Ένωση και είδαμε πώς ισχυροποιήθηκε η Ένωση και έτσι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η προσφυγική κρίση. Στο Πανεπιστήμιο μου δόθηκε μια υποτροφία για να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες στο εξωτερικό και ήταν μια ευκαιρία την οποία δεν θα είχα χωρίς την οικονομική και πανεπιστημιακή στήριξη της Ένωσης. Οπότε έμαθα από πρώτο χέρι το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή των νέων. Ανεξαρτήτως ε, από πού προέρχονται. Τον ε, Νοέμβριο έφερα την εκστρατεία των φιλελεύθερων σε υπεράσμους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε τώρα 10.000 υποστηρικτές ε, και ο κάθε ένας από αυτούς έχει μια μοναδική εμπειρία για το πώς άλλαξε η ζωή τους με τις ανταλλαγές αυτές. Κάποιοι από αυτούς που ανησυχούν περισσότερα ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν 17 ετών, δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα, αλλά γνωρίζουν ότι απειλούνται οι μελλοντικέ ευκαιρίες τους. Εμείς λοιπόν δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί θεατές, ενώ η Βρετανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται την μελλοντική μας ε, θέση. Θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι ανταλλαγές και η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus Plus. Ελπίζουμε οι ευρωβουλευτές και τα μέλη της ε, Κομισιόν να μας υποστηρίξουν στο να αποκτήσουμε το καθεστώς χώρας, ε, τρίτης χώρας η οποία συμμετέχει. Έτσι θα μπορούμε να σπουδάζουμε στο εξωτερικό και οι νέοι Βρετανοί θα είναι κάτι το οποίο ελπίζω να σας απασχολεί στις διαπραγματεύσεις. Να θυμάστε ότι οι περισσότεροι από μας ψηφίσαμε να μείνουμε στην Ένωση. Όταν η Τερέζα Μέη προκήρυξε πρόορες εκλογές, όπως είπατε περίμενε να ενισχυθεί η θέση της, αλλά οι Βρετανοί έδειξαν ότι δεν ήθελαν αυτήν την προσέγγιση στο Brexit και άρα έχασε την αυτοδυναμία στο Κοινοβούλιο και εγώ είμαι υπερήφανη που ανήκω στους ε, φιλελεύθερους ε, δημοκράτες. Θεωρούμε ότι το Brexit είναι ένα τεράστιο λάθος ε, και κάποια στιγμή όταν αναγνωριστεί αυτό ελπίζουμε οι νέοι να επαναφέρουν το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να καταστεί αυτό δυνατόν πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να αναπτυσσόμαστε μαζί με τους Ευρωπαίους γειτονές μας. Γι' αυτό ζητάμε να μας στηρίξετε στην εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Και τώρα θα σας δείξω κάποια μέλη της εκστρατείας μας στο βίντεο. Um, it wasn't what I'd wanted and what the other young people had wanted. Uh, and uh, I felt that the voting age should have been lowered in that case. You know,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 Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε την ε, κάμερα αυτή που είναι στο διαδίκτυο και δεν είδατε αυτό το οποίο είδα εγώ, τα, τα πρόσωπα. Θεωρώ ότι και Όσκαρ να έπαιρναν δεν θα έκαναν έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή είναι η δύναμη της ευρωπαϊκής ιδέας. Έχουμε ολόκληρη την Βρετανική κοινωνία που μας λέει ότι θέλει να παραμείνει και σας ευχαριστώ πραγματικά σας είμαι ευγνώμων. Εννοείται ότι θα παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Θα στείλουμε ως προτεραιότητα στην Κομισιόν και όλοι, όλοι θα δουν αυτό το βίντεο, θα το λάβουν τουλάχιστον όλοι οι ευρωβουλευτές. Λοιπόν, αυτή ήταν η τελευταία ακρόαση για το Brexit. Κυρίες και κύριοι, και τώρα έχουμε την 952 ε, την 832-16 την 872 την 1225 ε, την 352 ε, την 787 και την 788 του 16 είναι στην Κομισιόν και τώρα περνάμε στο τελευταίο θέμα της ε, σημερινής ημέρας ε, η συνάδος Ήβη θα μας πει για μια γνώμοδότηση Έχετε λοιπόν τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε προς η συγγετρία. Σχετικά με την Πρώτα επαφορά αφορά ΑΠΕ να τονίσω ότι η γραμματότηση αυτή χαρακτηρίζεται από την βούληση αξιοποίησης των πολιτών και των οργανώσεων πολιτών όσον αφορά την παραγωγή και χρήση των ΑΠΕ, δίνοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες απαντήσεις στις ανησυχίες των πολιτών μέσω των αναφορών που έχουμε δεχτεί εδώ στην Επιτροπή μας. Να σας πω αμέσως ότι κάποια τεχνικά ζητήματα προτίμησα να τα παραπέμψω σε άλλες αρμόδιες επιτροπές όπως αυτή για το περιβάλλον και την ενέργεια. Η γνωμοδότηση που παρουσιάζω επικεντρώνεται σε ένα σύνολο τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθώντας να κάνουμε το πλαίσιο αυτό όσο πιο φιλόδοξο γίνεται. Καταρχάς όσον αφορά τους στόχους για τις ΑΠΕ το 2030. Και αυτό το λέω για ένα απλό λόγο. Το 2050 να έχουμε 100% ΑΠΕ. Στόχος φιλόδοξος που ήδη από σήμερα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται. Πετυχαίνοντας ένα διάμεσο στόχο όπως αυτό αυτούς του 2030. Οι μελέτες που διαθέτουμε μας λένε ότι οι ΑΠΕ στην Ένωση, αν αξιοποιηθούν σωστά και στηριχτούν από ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο, μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός στόχου της τάξης του 45% το 2030 και αυτό το στόχο 45% θέλησε να περιληφθεί εδώ στην ε, νομοδότηση. Η Κομισιόν ως το 2020 έχει ως στόχο το 20% των ΑΠΕ. Κάτι που φαίνεται να μπορούν να πετύχουν είναι οι χώρες της Ένωσης. Ο νέος στόχος όμως για το 30-45% ετησίως αντιπροσωπεύει μια αύξηση 2,5%. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο σωστός δρόμος για να καταλήξουμε στο 100% το 2050. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι να αποδεχτούμε το ανεπαρκές 27% που ανταποκρίνεται ή αντιστοιχεί σε μια αύξηση με 10,7% μέχρι 2030. αφήνοντας ένα δύσκολο να εκπληρωθεί στόχο μετά το 2030. Από τις ίδιες τις μελέτες της Κομισιόν, αν η Ευρώπη σήμερα δεν κάνει τίποτα και συνεχίσει να κάνει αυτά που κάνει, το 2030 θα είχε φτάσει στο 24,3%. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω, για να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Πέραν των στόχων, σκεφτήκαμε να επαναθέσουμε στόχους δεσμευτικούς σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο ενωσιακούς στόχους δηλαδή. Και πάλι η ίδια η Κομισιόν στη δική της την αξιολόγηση στα πλαίσια του ΡΕΦΗ το Νοέμβριο του 2016 είπε ότι η εθνικοί στόχοι, οι δεσμευτικοί, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη πολιτικών και επενδύσεων για τις απέστης χώρες μέλη. Σε αυτή λοιπόν την γνωμοδότηση θέλησα επίση να αντιμετωπίσω ή να προσεγγίσω ένα άλλο ζήτημα που θίγουν διάφορε αναφορέ, δηλαδή η σταθερότητα του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις ΑΠΕ. Συχνά είδαμε αναδρομικές νομοθετικές αλλαγές ή κανονιστικά πλαίσια ασταθή και διαφανή κάτι το οποίο δεν βοήθησε την διάδοση των ΑΠΕ. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε προς μια μεγαλύτερη σταθερότητα όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό επειδή οι κίνδυνοι σχετικά με τις επενδύσεις στον κλάδο αυτό έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Και πολλές αναφορές κατέδειξαν ακριβώς την έλλειψη εμπιστοσύνη εκ των πολιτών για τα σχέδια που αφορούν ΑΠΕ. Ακριβώς λόγω αναδρομικών τροποποιήσεων στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Γνωστό παράδειγμα η Ισπανία, για το οποίο έχουμε δεχτεί πολλές ε, αναφορές και αφορούν τα φωτοβολταϊκά. Νομίζω ότι οι μόνες τροποποιήσεις που θα μπορούσαμε να προβλέψουμε είναι αυτές που αφορούν μόνο στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, ώστε αυτή να είναι περιεκτική και διαφανής, χωρίς τροποποίησεις αναδρομικές. Προσωπικά να πω ότι η ενεργειακή μετάβαση στις ΑΠΕ σημαίνει ότι στοχεύουμε σε ένα σύστημα ενέργειας το οποίο αποβλέπει σε ωφέλη για όλη την κοινωνία, ώστε να καταστήσουμε δημοκρατικό το ενεργειακό σύστημα και όσο γίνεται αποκεντρωμένο. Σήμερα πραγματικά ζούμε σε μια κατάσταση όπου ελάχιστοι όμιλοι κατέχουν την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας. Πρέπει να αντιστραφεί αυτό το μοντέλο, ώστε να καταστεί δημοκρατική ενέργεια. Ο ρόλος των πολιτών, των καταναλωτών, των κοινοτήτων που παράγουν και καταναλώνουν ενέργειες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Και πράγματι έτσι θα πρέπει να ειδωθεί ο ορισμός που προσέθεσα τον απέως κοινό αγαθό. Γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε κίνητρα και οικονομικά στους prosumer, τους αυτοπαραγωγούς στον χώρο των ΑΠΕ. Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να προσεγγίσουμε μέσω των πολιτικών για τις ΑΠΕ είναι η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Γιατί δυστυχώ 11% μας λένε οι επίσημες στατιστικές, 11% πλήττεται ή κινδυνεύει από ενεργειακή φτώχεια. Εδώ λοιπόν οι πολιτικές των ΑΠΕ θα μπορούσαν να παράσχουν μεγάλε ευκαιρίε για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Ένα άλλο ζήτημα που θέλησα να προσεγγίσω σε αυτή τη γνωμοδότηση αφορά κάτι άλλο που θέλησε να αφαιρέσει η Κομισιόν από αυτή την πρόταση τροποποίηση που θέλησα εγώ να επαναφέρω γιατί η αναδιανομή και η δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο ενέργειας που παράγουν ΑΠΕ ήταν ένα αποτέλεσμα θετικό που μπορούσαμε να δούμε στο σχεδιασμό των προγραμμάτων για τις ΑΠΕ σε εθνικό επίπεδο. Και τέλος, να μην κρύβουμε το εξής, ότι άμεσες ή έμεσες ενισχύσεις εθνικές προς τις ΑΠΕ από ρηκτά καύσιμα. Υπάρχουν ακόμα και θα πρέπει να αρθούν, να εξαλειφθούν οι άμεσες ή έμεσες εθνικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις των ρηκτών καυσίμων αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ενεργειακή μετάβαση και να προωθήσουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αυτές είναι οι προτάσεις μου στα πλαίσια της νομοδότησης. Θα καλοποιήσω βέβαια περαιτέρω στο κείμενο με τις τροπολογίες να αναφερθώ σε μία συγκεκριμένα, να συμφωνήσουμε δηλαδή για το τι θεωρούμε ή τι εννοούμε με ενεργειακή ανάκτηση των απορριμμάτων. Η αποτέφρωση είναι μία πρακτική που είναι διαδεδομένη και επιδοτείται υπερβολικά. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτές τις κρατικές επιδοτήσεις που αφορούν την ενεργειακή ανάκτηση και αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων. Όπως εξάλλου είπε και η, η ανέξη της Κομισιόν που ακριβώς για αυτό το πράγμα μιλάει, για την κατάψη αυτών των πρακτικών δηλαδή, εκ μέρους των χωρών Αυτά από μένα, ευχαριστώ και προσμένω τα σχόλιά σας και προσβλέπω σε θετική συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε τον λόγο. Ε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρόσκη μου ζήτησε να μεταφέρω τα σχολεία της. Και θα πέρασω στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της που έχει κάνει. Η γνωμοδότηση λαμβάνει υπόψη κάποια πάρα πολύ σημαντικά σημεία που επηρεάζουν του Ευρωπαίου πολίτε όμω δεν εστιάζει αρκετά στι αναφορέ που έχουμε λάβει. Πρέπει να δώσουμε περισσότερο πάρο στι αναφορέ και να εστιαστούμε συγκεκριμένες ανησυχίες. Αυτό έχει συμφωνηθεί και στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιτροπών και θα υποβάλω τις ανάλογες ε, τροπολογίες. Μία από τις κύριες ε, πτυχές αφορά την περισσότερη νομική βεβαιότητα στις επενδύσεις της ΑΠΕ. Πολλοί καταναλωτές διστάζουν να επενδύσουν λόγω της αβεβαιότητας διαφόρων νομικών καθιστώτων στα 28 κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν ε, διαφορετικά καθιστώτα επιδοτήσεων στα κράτη-μέλη και δεν πρέπει να αγνοούμε τι αναφορέ των Ευρωπαίων πολιτών. Η επιθυμία για διαφάνεια και σταθερότητα φαίνεται και στι αναφορέ που λάβαμε τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, πολλοί αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία του όταν μιλάμε για την διάρκεια των εγγυήσεων επενδύσεων σε ΑΠΕ. Μια αλλαγή κυβέρνησης ε, δεν πρέπει να σημαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που έχουν ήδη δοθεί μπορούν να χαθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριος Γιάρ. Ναι. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια για τις παρατηρήσεις της. Χαμόγελασα λίγο κάπου και όπου είπε η κυρία Εύη ότι δεν πρέπει να γίνεται πλέον καύση των απορριμμάτων ε, είναι πάρα πολύ κακό. Είχα πάει όμως σε μία επίσκεψη στην Ιταλία και πρέπει να σας πω ανοιχτά ε, βλέπουμε ανοιχτές χωματερές ε, παντού, δηλαδή μακάρι να υπήρχε οργανωμένη καύση. Εντάξει, ωραίο είναι να τα λέμε αυτά, αλλά μην ξεχνάμε για την πραγματικότητα που υπάρχει. Και όταν υπερβάλλουμε, καμιά φορά δεν αξίζουν τα πράγματα που λέμε, ούτε το χαρτί στο οποίο τα γράφουμε. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό τώρα. Αυτά ήταν στην ευρύτερη περιοχή της, ε, της Νάπολης. Ε, αν είχαμε εγκαταστάσεις απανθράκωσης δεν θα είχαμε όλα αυτά τα ωραία που είδαμε εκεί. Λοιπόν, το είπαν οι προλαλήσαντες, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών και πρέπει οπωσδήποτε να μην βλέπουμε σε αρμοδιότητες άλλων επιτροπών. Δηλαδή πρέπει να προσανατολισόμαστε στις αναφορές που υπάρχουν και ανάλογα να τοποθετηθούμε. Αυτό έχει δύο επιδράσεις ότι θα πρέπει να είμαστε ε, σύντομοι και να λέμε και πράγματα πιο ουσιαστικά. Έτσι θα μας πάρουν και πιο σοβαρά οι άλλες επιτροπές. Ανέφερε και συνάδελφος από τους σοσιαλδημοκράτες κάποια καλά παραδείγματα του τι μπορεί να γίνει. Και τα οποία μπορούμε να υποβάλουμε ως ε, τροπολογίες. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε τους στόχους. Έχουμε... Ναι, η δικιά μου η ομάδα θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρχουν πανευρωπαϊκοί στόχοι και βέβαια θεωρούμε σωστό να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και απαραίτητη βεβαιότητα για να γίνουν οι επενδύσεις. Για το θέμα των αυτοπαραγωγών ε, τώρα ΑΠΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη βεβαίως πρέπει να προσέξουμε να μην ε, φύγουμε από τη μία παχύδα και πέσουμε στην άλλη μέσω των θετικών λεγόμενων ε, διακρίσεων. Αυτά θα υποβάλουμε και τις ανάλογες τροπολογίες οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ. Ε, τώρα έφτασε η ώρα να θέσουμε μια ερώτηση στην Κομισιόν. Ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει με χαρά το ενδιαφέρον να αναθεωρηθεί η νέα ε, οδηγία για την ενέργεια. Αυτό Βάνοντα υπόψη ότι υπάρχουν πολλές επιτροπές, πάνω από 7 επιτροπές ε, που είναι συνδεδεμένε με αυτή την πρόταση. Η πρόταση είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ε, επιτύχουν ε, τον στόχο για τι ανανεώσιμε μέχρι το 2030. Και αυτό λοιπόν είναι προτεραιότητα της Ένωσης να γίνει η νούμερο ένα στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι καταναλωτές να μπουν στο κέντρο της Ενεργειακής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζει και η συγγήτρια. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά το στόχο. Η πρότασή μας στηρίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ξεπερνά ε, την απλή δημιουργία ενός στόχου. Δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ασφάλειες επενδύσεις, για ε, ασφάλεια των ε, καταναλωτών και προτείνει φιλόδοξα μέτρα σε πολλούς τομείς, την ψήξη, θέρμανση, ηλεκτρισμό και τις μεταφορές έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό των ανανεώσιμων. Όλο αυτό θα γίνει σε συνδυασμό με την ε, πρόταση της θέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια όλους τους Ευρωπαίους. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι μετά από αυτά μπορούμε να ε, δούμε μια πρόταση που θα ευδοκιμήσει. Η πρόταση της εισηγήτριας ε, είναι ε, μια πρόταση που συμφωνεί και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως είναι η τιμές υψηλότερες από ε, την πρόταση της Επιτροπής Ήτρε και το 30% των προηγούμενων ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης συμφωνεί απόλυτα με κάτι που ε, εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές, δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη σταθερού ε, ρυθμιστικού πλαισίου. Γι' αυτό προτείνουμε αρκετά άρθρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επενδυτών. Το άρθρο 6 είναι ένα από αυτά, όπου υπάρχει μία διάταξη για να ε, αποφύγουμε την αναθεώρηση των διάφορων ε, προγραμμάτων στήριξης και να κινδυνεύσει λοιπόν η χρηματοδότηση πολλών έργων. Σε ό,τι αφορά τους ε, καταναλωτές που παράγουν ίδια ενέργεια και τις ενεργειακές κοινότητες, να πω πως μία από τις προτεραιότητές μας είναι οι καταναλωτές να μπουν στο κέντρο της Ενεργειακής Ένωσης, επαναλαμβάνω, και για πρώτη φορά δημιουργούμε το δικαίωμα της αυτοκατανάλωσης, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να το ασκήσει. Πιστεύουμε πως η πρότασή μας παρέχει πολλές καλές ευκαιρίες για τους καταναλωτές και για τις ε, ενεργειακές κοινότητες, διατηρώντας επίσης την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ενέργειας. Από την άλλη όμως, πιστεύουμε ότι έχουμε μια αρκετά ισορροπημένη προσέγγιση έτσι ώστε οι καταναλωτές παράγουν μόνοι τους ενέργεια να μην ε, επιβαρύνουν το σύστημα, αλλά να συνεισφέρουν σε αυτό. Και σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση για πρόσβαση προτεραιότητας ε, στη δυναμία, να πω ότι η οδηγία για τις ε, ανανεώσιμες διαγράφει το σημείο αυτό. Διότι αυτό έχει μεταφερθεί σε άλλο κομμάτι νομοθεσίας, στον κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια. Δεν εξαφανίστηκε λοιπόν, δεν διαγράφηκε, μεταφέρθηκε με κάποιες τροποποίησεις αλλού. Θα ήθελα εδώ λοιπόν να καλέσω το Κοινοβούλιο να υποβάλει τις τροπολογίες του για αυτό το θέμα, για τον κανονισμό, έτσι ώστε να μην ε, υπάρχουν ε, επαναλήψεις σε άλλα ε, νομοθετήματα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ορυκτά καύσιμα που βασίζονται σε απορρίμματα. Φαίνεται πως εδώ υπάρχουν διάφορα θέματα που γύρουν πολλά ερωτηματικά και θα ήθελα να πω ότι αυτό, αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό της ανανεώσιμης ενέργειας, δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν προσμετρώνται στους στόχους ανανεώσιμων μόνο στις υποχρεώσεις των ε, επιχείρησεων σχετικά με τους προμηθευτές και τη μεταφορά καυσίμων ε, και στους ε, στόχους για απεξάρτηση από τον άνθρακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. καταληκτική ημερομηνία υποβολή τροπολογιών 29 Ιουνίου, 3 το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Αναφορών στις 7 Σεπτεμβρίου. Κυρία Εύη, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι? Ευχαριστώ στους αδελφού. Θα συνεργαστούμε νομίζω, γιατί αυτά που είπατε κι εσείς εν μέρει τα αναφέρω και εγώ στη γνωμοδότηση. Όπως υπενθύμησαν δύο συνάδελφοι και από τις πολλές αναφορές, αυτά που είπατε θα αποτελέσουν το επίκεντρο της νομοδότησης. Όπως και αυτά είπαμε για τους στόχους. Ελπίζω το κείμενο να έχει φιλόδοξη θέση στο Κοινοβούλιο γιατί ξέρουμε μετά, τα έχουμε διαπραγματεύσει και τριμερεί διαλόγου με το Συμβούλιο και συχνά χάνουμε αυτή τη φιλοδοξία. Οπότε με τις προσπαθειές μας ελπίζουμε να έχουμε μακρόπνοες ε, πολιτικές υπέρ του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 το πρωί και σας εύχομαι καλό βράδυ.